Πρόεδρο. thought so. Okay, colleagues. Πρόεδρος, αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε ωραία και τακτικά. Έχουμε εδώ δύο προεδρεύοντες εκπροσωπούντες την ελληνική προεδρία. γιατί οι Έλληνες φυσικά έχουν ε, ξεχωριστό Υπουργείο Ναυτιλίας που αν δεν είναι ασφαλό ονομάζεται Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου με Υπουργό τον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη ο οποίος θα μιλήσει και πρώτος. Μετά έχουμε και τον ε, κύριο Χρυσοχοίδη λέει ο πρόεδρος εξ ονόματος του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων θα δώσω πρώτα τον λόγο στον κύριο Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος είναι Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου και θα μας μιλήσει εξ ονόματος της Ελληνικής Προεδρίας. Πιστεύω ότι έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά τις ολοκληρώσατε μετά με διδακτορικές σπουδές στο Χάρβαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι μεγάλη χαρά για μένα να είμαι εδώ παρόν με εσά. Όπω ξέρετε, η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου σε μια συγκυρία όπου λόγω τη χρηματοπιστωτική κρίση, αλλά κρίσιμη συγκυρία και για τι εργασίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διότι έχουμε μόνο ε, μισό εξάμεινο γιατί κατόπιν στα μέσα της Προεδρίας μας ε, το Κοινοβούλιο θα διαλυθεί. Άρα πρέπει να βιαστούμε για να λύσουμε τα εκκρεμή θέματα, αλλά πολλά έχουν ήδη προωθηθεί τα τελευταία χρόνια και κατά πάσα πιθανότητα θα είμαστε σε θέση να δρέψουμε κάποιους καρπούς από τη συνεργασία μας. Πρώτα απ' όλα προσωπικά αλλά και ως Προεδρία προσβλέπουμε στη συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Και πιστεύουμε ότι η εργασία που κάνει το Κοινοβούλιο και οι παρατηρήσεις που κάνουν οι ευρωβουλευτές για την νομοθεσία ή που εκπώνηση είναι πολύ σημαντική για την Προεδρία για να ε, επιτευχθούν κοινέ θέσει στο Συμβουλίο. Οι παρατηρήσεις των βουλευτών πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη σοβαρά γιατί είναι έκφραση των διαφόρων συζητήσεων και διαφορετικών απόψεων για θέματα που είναι επίμαχα. Καταρχάς, να πω λίγα λόγια για το γιατί θα υπάρχουν δύο προεδρεύοντες σε σχέση με την Επιτροπή σας από τη μία με εγώ και από την άλλη ο κύριος Χρυσοκοίδη. Θα είμαστε συμπρόεδροι. Όπως ξέρετε, παραδοσιακά η Ελλάδα είναι ναυτική χώρα. Εξαρτώμεθα από τη θάλασσα για την οικονομική μας ανάπτυξη αλλά και για τον ε, πολιτισμό μας. Ο πολιτισμός μας έχει μεγάλη σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον. Γι' αυτό Υπάρχει ε, ειδικευμένο Υπουργείο για τα θέματα θάλασσας αλλά και ναυτιλίας. Γιατί και η ναυτιλία είναι πολύ σημαντική και για την ευρωπαϊκή και, την παγκόσμια, και την ευρωπαϊκή οικονομία. Το θαλάσσιο εμπόριο είναι 98% του ευρωπαϊκού εμπόριου. Περίπου όλα τα ενεργειακά μας προϊόντα φτάνουν ε, μέσω θαλάσσης και το μεγαλύτερο τμήμα των εισαγωγών-εξαγωγών μας γίνεται μέσω θαλάσσης. Ως Ελλάδα έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς στόλους. Είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερα την αυτιλία και το εμπόριο. Το ελληνικό νεολόγιο έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 1500 ε, σκάφη και αποτελεί πάνω από 40% του ευρωπαϊκού στόλου και 15% του παγκόσμιου στόλου. Και επειδή είμαστε λοιπόν σημαντικός ε, διεθνής παράγοντας στην αυτιλία, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για το εμπόριο μέσω θαλάσσης και θέλουμε να εστιάσουμε και να στείλουμε ένα μήνυμα σε όλη την Ευρώπη και στο Κοινοβούλιο. Το εξή μήνυμα. Η ναυτιλία, ο κλάδος της ναυτιλίας δεν θα πρέπει να μεταφερθεί σε άλλα μέρη του κόσμου. Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας ε, της ευρωπαϊκής ναυτιλίας είναι πρωταρχικής σημασίας. Η Ευρώπη συνολικά κερδίζει από το να είναι νεολογημένα τα πλοία εδώ, να έχουν την έδρα τους ναυτιλιακές εταιρείε, τα καράβια που διασχίζουν τους ωκεανούς και παρέχουν ναυτιλιακές υπηρεσίες να έχουν ευρωπαϊκές σημαίες. Δεν θα πρέπει να προωθήσουμε περιφερειακές πολιτικές που θα διώξουν όχι μόνο από τη χώρα μου αλλά και από άλλες χώρες που έχουν ναυτιλία θα διώξουν λοιπόν εκτός Ευρώπης ένα μεγάλο τμήμα του ναυτιλιακού κλάδου. Είναι ζωτική σημασία για την Ένωση να παραμείνει η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη παγκόσμια. Πρέπει λοιπόν να διατηρήσουμε το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα για την Προεδρία μας, ένα από τα θέματα κλειδιά, ένας από τους πυλώνες που θέτουμε ως προτεραιότητα της Προεδρίας μας είναι ο πυλώνας θάλασσα. Είναι και οικονομικό θέμα ενίσχυση της Ευρωζώνης. Επίσης θέλουμε ανάπτυξη και απασχόληση. Ένας τρίτος πυλώνας ε, αφορά την μετανάστευση. Και ο τέταρτος πυλώνας της Προεδρίας μας είναι ο πυλώνας που αποκαλούμε θάλασσα. Διότι η μπλε οικονομία, η γαλάζια οικονομία έχει τεράστια δυνατότητα καινοτομίας, ανάπτυξης, ε, απασχόλησης. Η γαλάζια οικονομία αποτελεί αυτή τη στιγμή ε, δίνει 5,4 εκατομμύρια θέσεων εργασίας και περίπου 500 δισεκατομμύρια ε, ακαθάριστο εισόδημα ετησίως. Η οριζόντια θεματική μας λοιπόν που θα εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς προτεραιότητας και για την ανάπτυξη, για την απασχόληση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, ε, μετανάστευση και σύνορα και φυσικά η ναυτιλιακή πολιτική, η ολοκληρωμένη ναυτιλιακή πολιτική, η θαλάσσια πολιτική, οι μεταφορές, ε, η αντιμετώπιση του νησιωτικού χαρακτήρα, η μετανάστευση μέσω της θάλασσας και η ασφάλεια και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών μας. Όλα αυτά πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα τους επόμενους μήνες, ούτω ώστε να καταφανεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το τμήμα της οικονομίας μας, αλλά και της ε, κοινωνικής και εθνικής μας ανάπτυξης. Είναι πολύ σημαντικά αυτά που ήδη κάνατε. Ξέρω ότι ο κύριος Σίμψον έχει καταβάλει τεράστιες προσπάθειες για να αυξηθεί η ασφάλεια και προστασία στη θάλασσα. Αυτός ο νέος κανονισμός για τον ε, ναυτικό εξοπλισμό και ο κανονισμός υποεκπώνηση για άλλα θέματα κλειδιά που πρέπει να μας απασχολήσουν και για τα οποία πρέπει οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε κοινή στάση με την ε, Επιτροπή και το Συμβούλιο, ούτως ώστε να έχουμε καθαρές θάλασσες, τα σκάφη μας να έχουν σύγχρονο εξοπλισμό. Όλα αυτά είναι πρωταρχική σημασία για μια ναυτική χώρα, για μια χώρα που περιβρέχεται από, τόσα παράλια, από τόσες θάλασσες και έχει τόσα παράλια όπως εμείς και γι' αυτό θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο. Κάτι άλλο, στο οποίο θα στοχεύσουμε. Να ενισχυθεί η συνεργασία μας με τον Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Οργανισμό. Πιστεύουμε ότι οι διεθνείς σχέσεις, οι διεθνείς σχέσεις και αυτό είναι προτεραιότητα εντός του Συμβουλίου, οι διεθνείς σχέσεις στον τομέα της ναυτιλίας είναι σημαντικές. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούν στενότερα ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός με την Ένωση για να εκπονηθεί περαιτέρω ένα αριθμιστικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι οι ανοιχτέ θάλασσε και οι ανοιχτοί λιμένες είναι σημαντικό για την Ευρώπη, για μας, για την ναυτιλία. Ήδη λοιπόν πληροφορήσαμε την Κομισιόν ότι θα καλέσουμε το Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας να συμμετάσχει στην έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου το Μάιο στην Αθήνα για να ενταθεί η συνεργασία για τα θέματα αυτά. Τώρα, τι νομοθετικές προτάσεις έχουμε για την αυτιλία. Θέλουμε να σημειωθεί πρόοδος για να καταλήξουν οι συζητήσεις σε πρώτη ανάγνωση για μια σειρά προτάσεις στις οποίες θα αναφερθώ. Πρώτον, όπως ήδη είπα, με την ε, στήριξή σας θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία για την οδηγία για τον ε, ναυτιλιακό εξοπλισμό σε πρώτη ανάγνωση του ώστε μέσω της έγκρισης της πρότασης αυτής να ενισχυθεί ε, ο μηχανισμός εφαρμογής και να ελέγξουμε τις προποθέσει για τον ε, εξοπλισμό των πλοίων, την ε, απλοποίηση των κανόνων, ούτω ώστε να είμαστε σίγουροι ότι οι απαιτήσει του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού θα εφαρμοστούν με εναρμονισμένο τρόπο από τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την πρόταση κανονισμού για την πολιετή χρηματοδότηση, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα στον τομέα τη αντιμετώπιση τη μόλυνση που προκαλείται από τα πλοία και τη θαλάσσια μόλυνση που προκαλείται από εγκαταστάσει πετρελαίου και φυσικού αερίου θα προσπαθήσουμε να υπάρξει συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην πρώτη ανάγνωση. Υπογραμμίζω ότι η Ελληνική Προεδρία αναγνωρίζει την αναγκαιότητα να υπάρχει οικονομική βιωσιμότητα του Ευρωπαϊκού ε, Ναυτιλιακού Οργανισμού για ασφάλεια στη θάλασσα για να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση στη θάλασσα. Θα κάνουμε κάθε προσπάθεια για επιτυχή κατάληξη των ε, συζητήσεων. Όπως ε, είπα ήδη, η Ελληνική Προεδρία αντιλαμβάνεται την ανάγκη για να δημιουργηθεί πιο ευνοϊκό περιβάλλον για επενδύσεις στους λιμένες. Θα επιτύχουμε λοιπόν να υπάρξει πρόοδο στο Συμβούλιο για την πρόταση κανονισμού για να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο για, για ε, να μην υπάρχουν διακρίσεις στην πρόσβαση στις λιμενικές υπηρεσίες και την ε, οικονομική διαφάνεια των λιμένων. Επίσης υπάρχει πολύ εκτεταμένο πρόγραμμα ιδιωτικοποίησης των λιμένων μας, γι' αυτό θέλουμε συγκεκριμένους κανόνες για τον τρόπο λειτουργίας των λιμένων μας. Αλλά ξέρω ότι ως βουλευτής, ξέρω ως βουλευτής που είμαι, ότι υπάρχουν ε, δύσκολα και επίμαχα θέματα γύρω από αυτό και ορισμένες φορές σε προεκλογική περίοδο είναι δύσκολο να καταλήξουν τέτοια συζητήσεις, αλλά ως Προεδρία θα επιδιώξουμε να ε, ε, καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση. Η Προεδρία αποδίδει πολιτική σημασία Στη διαδικασία εντό του Συμβουλίου με στόχο την εκπόνηση ενό νομοθετικού κειμένου που θα συμβάλλει στην ανάπτυξη, την απρόσκοπτη λειτουργία τη ενιαία αγορά και τη δημιουργία ενό σταθερού περιβάλλοντο, ούτω ώστε να μην υπάρχουν διακρίσει στα λιμάνια, σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη και τις άλλες, ε, τα άλλα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Όπως σας είπα, ήδη θα υπάρξει ένα άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ναυτιλίας αρχές Μαΐου στην Αθήνα στην οποία συνάντηση θα κάνουμε την, μέσο, ε, την ενδιάμεση αναθεώρηση της ε, ε, πολιτικής μας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Τέλος. Στα πλαίσια του Συμβουλίου θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα του νησιωτικού χαρακτήρα και του τουρισμού στα νησιά μαζί με τα αρμόδια υπουργεία. Είναι και αυτό σημαντικό στόχος της Προεδρίας μας. Και πρώτη απτή θα έλεγα προτεραιότητα στα πλαίσια της ολοκληρωμένης ε, θαλάσσιας πολιτικής είναι να καταλήξουν οι πραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο για την πρόταση οδηγίας για τη δημιουργία δικτύου και πλαισίου για την, ε, τον χωροταξικό σχεδιασμό στις θάλασσες και την αντιμετώπιση των θεμάτων ε, διαχείρισης των ε, ακτογραμμών και παραλίων. Θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στην πρώτη ανάγνωση. Θα προωθήσουμε τις πρωτοβουλίες της Κομισιόν για τη στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη και για βιώσιμη ανάπτυξη στο θαλάσσιο και ναυτικό τομέα που περιλαμβάνει λοιπόν το θαλάσσιο και παράκτιο τουρισμό, την γαλάζια ενέργεια, την καλλιέργεια και την αξιοποίηση των θαλάσσιων ορεικτών πόρων. Με βάση την διακήρυξη ορόσημο της ε, Λεμεσού θα προτείνουμε για το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2014 σχέδιο πορισμάτων για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, στο οποίο κείμενο θα περιέχονται κατευθύνσεις γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για πρωτοβουλίες στα πλαίσια της ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής και της γαλάζιας ανάπτυξης. Όπως σας είπα και στην αρχή, είμαι πεπισμένος ότι είναι μεν φιλόδοξο το πρόγραμμά μας, αλλά με τη στήριξή σας και την στενή συνεργασία και με τον Πρόεδρό σας θα έχουμε αυτά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν ε, τη στήριξή σας, τη βοήθειά σας, ούτως ώστε σε μια σύντομη περίοδο να επιτύχουμε τους στόχους μας και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη στήριξή σας μέχρι στιγμής και φυσικά προσλέπω στη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Κουμουτσάκος, ο κύριος Δανέλης, η κυρία Μάισνερ, ο κύριος Κράμερ, η κυρία Φώστερ, ο κύριος Στούσας και η κυρία Γκουρμάη έχουν εγγραφεί. Παρακαλώ να μην υπερβαίνετε τα τρία λεπτά έτσι ώστε και ο κύριος Υπουργό να έχει την δυνατότητα να απαντήσει σε ενδεχόμενες ερωτήσεις ή σχόλια που θα υποβάλλετε. Για τρία λεπτά ο κύριος Κουμουτσάκος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Μπράιαν. Κύριε Υπουργέ, σα καλωσορίζουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ιδιαίτερω δε στην Επιτροπή Μεταφορών. Σα ευχόμαστε τα καλύτερα για την ε, ελληνική Προεδρία. Ορθώ, αναφέρατε και υπογραμμίσατε μάλιστα ότι ε, η ναυτιλία, η ναυτιλιακή βιομηχανία και οι ε, θαλάσσιες μεταφορές σημαίνουν ανάπτυξη και θέσεις εργασίας και αναφερόμαστε δε στην, στα θέματα αυτά, η Ελλάδα οπωσδήποτε έχει ε, ένα λόγο να πει ε, και καταλαβαίνετε ότι ε, μάλιστα τη στιγμή που προεδρεύει η Ελλάδα στην Ευρώπη είναι ένας λόγος παραπάνω για να συζητήσει για τα θέματα αυτά που τόσο πολύ την ενδιαφέρουν. Αναφερθήκατε σε θέματα ε, νομοθεσίας, ε, θα τα αντιμετωπίσετε σε τέσσερις μήνες σχεδόν. Αυτό είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα φυσικά και ευελπιστώ ότι θα καταφέρετε να επιτύχετε όπως αναφέρατε και εσείς απτά αποτελέσματα. Θα ήθελα ως σκιώδης εισηγητής για τους λιμένες και για τον κανονισμό δηλαδή για τους λιμένες πρόσβαση ε, ε, και διαφάνεια όσον αφορά, οικονομική διαφάνεια όσον αφορά τους λιμένες. Θα ήθελα να πω το εξή. δεν ξέρω εάν αυτός ο κανονισμός έχει ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον, ε, αλλά είμαι βέβαιος ότι το παρελθόν του ήταν προβληματικό γιατί δεν καταφέραμε να επιτύχουμε κανονισμό. Είστε αισιόδοξο. Ποιο είναι το σχέδιό σας και το πρόγραμμά σας. Πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει κοινή προσέγγιση στους επόμενους 4-5 ε, μήνες. Ε, θα ήθελα να σας ε, επενέσω γιατί στην ατζέντα σας έχετε συμπεριλάβει και την στενή επαφή με τον IMO. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να αγνοήσουμε τον διεθνή τον Παγκόσμιο Οργανισμό ε, Ναυτιλίας, ε, τον IMO. Επίσης, ε, όσον αφορά την πρόταση οδηγίας για τον εξοπλισμό, είπατε ότι ευελπιστείτε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό είναι μάλλον φιλόδοξο ποια είναι τα σημεία, τα στοιχεία ή οι πληροφορίες που έχετε ε, που σας ε, ε, κάνουν να είστε αισιόδοξο. Ολοκληρώνοντας τις παρατηρήσεις μου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερα εξαντλητική και συνολική σας παρουσίαση. Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Κουμουτσάκο. Ο κύριος Δανέλης από την πλευρά των σοσιαλιστών είναι η αγαπημένη μου, έρχεται από την αγαπημένη μου πλευρά της Ελλάδας, από την Κρήτη. Κύριε Δανέλη, σας δίνω τον λόγο. Διπλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, αγαπητέ μου Υπουργέ, ε, θέλω να συγχαρώ την Ελληνική Προεδρία και να της ευχηθώ να ασκήσει το ρόλο της επικοδομητικά, αποτελεσματικά και να προωθήσει όσο το δυνατόν ε, την προστιλήση τους ζητήματα που αφορούν το κοινό μας σπίτι. Ε, και βεβαίως είναι απολύτως δεδομένο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα σταθεί επικοδομητικά στο πλάι της Προεδρίας για την επίτευξη όσο το δυνατόν περισσότερων ε, λύσεων στα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Θέλω να συγχαρώ την Προεδρία για την συμπερίληψη στις ε, προτεραιότητες της ε, γαλάζιας ανάπτυξης και συνολικά των ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την θαλάσσια οικονομία. Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε στο ότι ανοίγονται εξαιρετικές ευκαιρίες που θα ξανακάνουν ανταγωνιστική την Ένωση σε πολλούς από τους τομείς που ξέρει καλά ε, η Ευρώπη να χειρίζεται, το έχει αποδείξει αιώνες τώρα ε, και στον τομέα της παραγωγής πλούτου και στον τομέα της ε, δημιουργίας θέσεων εργασίας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω ποιες είναι οι τομεακές προτεραιότητες Προεδρίας σε σχέση με τη γαλάζια ανάπτυξη και τι είδους δράσεις σκοπεύετε να αναλάβετε. Και θέλω να σταθώ επίσης και σε ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη ε, των προοπτικών της γαλάζιας ανάπτυξης που δεν είναι άλλο από το εργαλείο του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Αναφερθήκατε, αυτό όμως που εισπράττουμε από το Συμβούλιο μιας και έχουν αρχίσει ήδη οι τρίλογοι είναι ότι ε, το Συμβούλιο δεν θέλει να, να, να, να φτάσουμε σε μια ουσιαστική οδηγία που θα δίνει λύσεις σε πολύ βασικά ζητήματα. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι όσο εντείνονται οι πιέσεις στη θάλασσα, όσο, όσο ανοίγονται νέοι τομείς, τόσο γίνεται και πιο επιτακτική η ανάγκη ε, μια συστηματικής και συντονισμένης και σχεδιασμένης διαχείρισης του θαλάσσιου και παρακτηριού χώρου σε όλα τα μέλη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε μια εικόνα του πώς σκοπεύετε εσείς ως Προεδρία να αντιμετωπίσετε επί της ουσίας αυτό και να μας δώσετε και μια ερμηνεία, αν είναι δυνατόν, γιατί η στάση του Συμβουλίου είναι τόσο ε, συντηρητική και ουσιαστικά ε, μπλοκάρει αυτή την εξέλιξη στον τομέα αυτό. Κλείνοντα, μια κουβέντα μονάχα για, τον, για τα λιμάνια, μια και έχουμε μπροστά, όπω και ο κ. Κουμουτσάκο ανέφερε, ένα, μια, ένα κρίσιμο ζήτημα. Ε, επειδή εμείς δεν έχουμε καταλήξει μια ομοφωνία σχετικά με τις ανεξάρτητες λιμενικές αρχές. Ε, η Προεδρία θα προωθήσει την ενσωμάτωσή τους στον ε, κανονισμό. Πώς σκέφτεται να το χειριστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Δανέλη. Κύριε Μάισνερ, μέρος των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Μια και ο Γιώργος Κουμουτζάκος, ο συνάδελφος, και έτσι Έλλην μίλησε στα αγγλικά, θα το πράξω και εγώ. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Κουμουτσάκος χωρίς μικρόφωνο δεν ακούστηκε. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι προερχόμενοι από μια εκλογική περιφέρεια με πολλούς λιμένες που βράχει η θάλασσα, είμαι και εγώ πολύ ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ναυτιλίας, είμαι υπεύθυνη για τις μεταφορές εκ μέρου των φιλελευθέρων, αλλά ιδιαίτερω με ενδιαφέρει η θάλασσα και σα ευγνωμονώ για αυτά που είπατε εδώ. Είμαι βεβαία ότι θα είναι σύντομη βεβαίω, όπως είπατε, η Προεδρία σας, μόνο τέσσερι μήνε, όπως είπατε, και είναι σύνομο και φιλόδοξη. Και είμαι βεβαία πολύ, πολλά θέματα νομοθετικά που έχετε ενώπιον σας, όπως και ο συναδελφό σας Υπουργός. Ε, μιλήσατε για την ε, θαλασσιά οικονομία και ανάπτυξη είναι ασφαλώς πυλώνας της Ευρώπης 2020 και της θετικής στρατηγικής. Προσφέρει πολλές δυνατότητες για πρόοδο. Έχουμε 40% του ΑΕΠ της Ευρώπης, ε, το οποίο παράγεται από την ναυτιλιακή οικονομία και θα αυξηθεί αυτό. Για να έχουμε λοιπόν αυτή την θαλασσιά οικονομία, νομίζω μπορούμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση και στην πολιτική για τους λιμένες. Όπως και ο Σπύρος Δανέλης θα ήθελα πιο πολλά πιο πολλές λεπτομέρειες, αν έχετε κάτι να μας δώσετε, για τις κατευθυντήριες γραμμές που ακολουθούν και τη διακήρυξη της, Λεμεσού, που ο Γιώργος, αν δεν απατώμε, και εγώ βεβαίως προσυπογράψαμε, ήμασταν παρόντες και περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα. Πακέτο για τους λιμένες ε, δεν θα σχολιάσω. Οδηγία για το θαλάσσιο εξοπλισμό θα είμαι εγώ εισηγήτρια και θα παρακολουθήσω τον διάλογο. Και για να ολοκληρώσω είμαι εισηγήτρια για τον ειδικό σχεδιασμό θαλασσών και για τη διαχείριση των ακτών. Κάναμε χθε μια πρώτη συνεδρίαση, πολλά υποσχόμενη συνάντηση και τη γνωρίζουμε το Συμβούλιο, τουλάχιστον κάποια κράτη-μέλη στο Συμβούλιο, είναι η υπήν διστακτικά. Δεν θέλουν να προχωρήσει η λύση. Εμεί πάντω το επιθυμούμε αυτό δεκώς και θεωρούμε ότι πρόκειται για μια αναγκαία επόμενη φάση, ένα επόμενο βήμα, να έχουμε το σχεδιασμό αυτών και να προχωρήσουμε. Και ξέρω ότι η Ελληνική Προεδρία ε, θέλει να βρει συμβαστικές λύσεις, θέλει να πείσει τους συναδέλφους της στο Συμβούλιο και σε αυτό θα ήθελα ιδιαίτερα να εκφράσω επενετικά λόγια. Έγινε λοιπόν, όπως είπα, μια πρώτη συνάντηση. Προσβλέπουμε στο προσεχή τριμερή διάλογο. Ευχαριστώ για τις προσπάθειές σας και για τα όσα κάνει η Ελλάδα για τι θάλασσες μεταφορές. Ευχαριστώ την κυρία Μάισνερ. Εκ μέρους των Πρασίμων, ο κύριο Κράμερ, Μάικλ. Εγώ πάλι θα μιλήσω τη μητρική μου γλώσσα, <laughs> τη γερμανική. Αλλά πρώτα θα σας πω Ευχαριστώ πολύ στα ελληνικά για την παρουσία σα εδώ και την ομιλία. Έχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχάς υπογραμμίζεται ότι η θαλάσσια οικονομία πρέπει να έχει μεγάλο μέλλον, ωστόσο υπάρχουν και σημεία επίκριση. Το είδαμε και στο θέμα των σιδηροδρόμων. Αν δεν επιληθεί το ζήτημα του θορύβου από του σιδηροδρόμου, παραμένουν τα προβλήματα. Το ίδιο και με τι θαλάσσιε μεταφορέ, οι οποίε δεν παρουσιάζουν στόχου μείωση και μέτρα μείωση ε, για τι ε, ζημιογόνε για το περιβάλλον εκπομπέ. Ξέρετε ότι έχουμε προϊόντα καύσεως από, τα, από το κατέργαστο πετρέλαιο που χρησιμοποιούν ως καύσιμο τα πλοία, που είναι πολύ επιβαρυντικά και ότι έχουν ε, συστήματα καύσεως χωρίς φίλτρο τα σκάφη. Τι βλέπετε λοιπόν σε αυτό και για το μέλλον, τι είδους δυνατότητες για περιορισμό των ζημιογόνων εκπομπών. Επίσης, μεταξύ Βόρειας και Βαλτικής θάλασσας είδαμε το 2005, από το 2005 σημαντική μείωση των εκπομπών θιούχων ενώσεων από τα σκάφη, αποτελέσματα που θα θέλαμε να γενικευθούν σε όλη την Ευρώπη. Ποια είναι η δική σας θέση. Βέβαια η Μεσόγειος έχει πλεονέκτημα ε, σε σχέση με τις βόρειες θάλασσες και ίσως τα προβλήματα και οι ρυθμίσεις αυτές να μην ισχύουν για τη Μεσόγειο. Βλέπετε κάποια σχέση ανταγωνισμού μεταξύ των ε, θαλασσών του Βορρά και της Μεσογείου ή παραμένει το πλεονέκτημα. Και κάτι ακόμα, η συζήτηση για την ε, οικονομική κρίση στην Ελλάδα που σοβεί ακόμη και στη Γερμανία μας λέει ότι υπάρχουν εκατομμυριούχοι της Ελλάδας, εφοπλιστές και είναι οι μόνοι οι οποίοι δεν πληρώνουν φόρο. Ο Υπουργό Εξωτερικών που είχε έρθει εδώ στι Βρυξέλλε ε, ε, κλήθη από τον υποφαινόμενο να απαντήσει σε μια σχετική ερώτηση και μου απάντησε ότι είναι τόσο περίπλοκο το θέμα που ακόμη το Σύνταγμα ορίζει ότι οι εφοπλιστέ εκατομμυριούχοι αυτοί, δισεκατομμυριούχοι αυτοί δεν πληρώνουν φόρο. Αυτό λοιπόν, δεδομένου ότι οι άλλοι όλοι οι εφοπλιστέ πληρώνουν φόρο σε άλλε χώρε, έχουμε να κάνουμε με θέμα τον ανταγωνισμό. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποιε είναι οι θέσει σα σε αυτό και βεβαίω για την ε, Μεσόγειο θέλουμε να δημιουργήσουμε όλοι όσο δυνατόν προσθέτει θέσει εργασία, αλλά πρέπει να εξασφαλίσουμε όχι μόνο την κινητικότητα αλλά και την προστασία του περιβάλλοντο. Και γι' αυτό θα ήθελα να μου πείτε σε σχέση με τι ε, πλωτέ συγκοινωνίε τη Μεσογείου, τι θέσεις έχετε. Ευχαριστώ κύριε Φώστερ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε. Όσον αφορά τις, ε, τους ε, φόρους ε, και το κατά πόσο πληρώνουν οι εφοπλιστές ή όχι. Αυτό είναι θέμα της ελληνικής κυβερνήσεως. Έχουμε άλλα θέματα να συζητήσουμε εδώ. Είμαι πολύ ευτυχής που αναφερθήκατε σε όλα αυτά τα θέματα. Είμαστε κι εμείς ναυτικό έθνος, το Ηνωμένο Βασίλειο, και ξέρουμε ότι ο, ο τομέας της ναυτιλίας και όσον αφορά την εμπορική ναυτιλία και όσον αφορά και τις κρουαζιέρες είναι πολύ σημαντικός τομέας για σας. Έκανα μια κρουαζιέρα μάλιστα στα ελληνικά νησιά, ήταν πολύ ευχάριστη. Τώρα πιο σοβαρά ε, φαντάζομαι ότι θα μιλήσετε και σε άλλες ε, επιτροπές ε, Βεβαίως το θέμα της μετανάστευσης είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βλέποντας τα θαλάσσια σύνορα, λαμβάνοντας υπόψη τις τραγωδίες τις οποίες είδαμε τα τελευταία χρόνια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία και σε άλλες χώρες, πραγματικά μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι κάτι πρέπει να γίνει. Δεν είναι δυνατόν ε, να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και βεβαίως δεν αφορά μονάχα την Επιτροπή Μεταφορών. Όσον αφορά τις υπηρεσίες θα ήθελα να πω ότι ε, εμείς στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, έχουμε ιδιωτικοποιήσει, έχουμε απελευθερώσει τα λιμάνια πριν από πάρα πολλά χρόνια με πολύ καλά αποτελέσματα. Η ιδιωτικοποίηση έδωσε πολύ καλά αποτελέσματα. Το θέμα είναι να γίνει με σωστό τρόπο στις διάφορες χώρες μέλη. Βεβαίως δεν πρόκειται να στηρίξουμε κάτι το οποίο θα αποβεί προς ζημίαν όλων των ε, οικοδομημάτων αν θέλετε και των επιτευγμάτων που έχουμε ε, μέχρι τώρα. Και δεν αναφέρομαι μονάχα στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες έχουν ε, ξεκινήσει, έχουν κάνει τα, τα βήματα αυτά και είμαι φανατικά υπέρ αυτής της κίνησης. Επίσης, όσον αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό και την διαχείριση των ακτών, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν μπορεί να έχουμε one size fits all, δεν μπορεί να είναι μία λύση που να ισχύει για όλους. Ε, θα πρέπει να δούμε οπωσδήποτε και την επικουρικότητα, θα πρέπει να δούμε ε, και να λάβουμε υπόψη τις ε, τοπικές ευαισθησίες, θα πρέπει να συζητηθούν τα θέματα με τα κράτη-μέλη, έτσι να δούμε ακριβώς πώς έχει η κατάσταση. Τέλος, ο ευθώς αναφερθήκατε στο ζήτημα του ε, IMO. Ε, ε, πιστεύουμε ότι το θέμα των, της, της θάλασσας, το θέμα, τα θέματα τα ναυτιλιακά ξεπερνούν αν θέλετε την Ευρώπη. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έρθουμε σε επαφή και να συμμορφούμε στα, και προς τις αποφάσεις του IMO. Θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και πρόσβαση στην τεχνογνωσία τους γιατί ασχολούνται και πάρα πολλά ε, χρόνια, δεκαετίες ε, με όλα τα θέματα αυτά. Επομένως ε, πιστεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να οδηγηθούμε σε σωστές λύσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στην Προεδρία σας και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τουσα. Έχετε τρία λεπτά κύριε Τούσα. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Τούσας. Πρέπει να ανοίξει το μικρόφωνο του. Sorry. Η γαλάζια ανάπτυξη, η ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, ενταγμένη στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ευρώπη 2020, προσφέρει ένα προνομιακό προκλητικά νομοθετικό πλαίσιο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της κερδοφορίας των εφοπλιστών και των μεγάλων επιχειρηματικών ομήλων στις θαλάσσιες μεταφορές αλλά και γενικότερα σε συνδυασμένες μεταφορές ακόμα και σε περίοδο κρίσης. Στοιχείο πρόχειρο που έχω είναι το εξή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του αφιλιακού τύπου αλλά και των οικονομικών εφημερίδων. Οι Έλληνες εφοπλιστές το 2013 επένδυσαν 18,2 δισεκατομμύρια ευρώ για την αγορά νεότευτων πλοίων και την ε, αγορά ε, δεύτερο χέρι πλοίων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις τράπεζές της ε, προσφέρει ένα μεγάλο κομμάτι που ξεπερνάει το 50% των επενδύσεων στην αυτιλία. Προσφέρει τις υποδομές, εξειδικευμένο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό, τις θέσεις των χωρών στους διεθνείς οργανισμούς και στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Δεν υιοθετώ σε καμία περίπτωση, είμαι ριζικά αντίθετος, ότι οι εφοπλιστές και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά τώρα και τα επόμενα χρόνια, μπορούν ανα πάσα στιγμή να πάρουν τα πλοία τους και να φύγουν. Ήδη έχει αλλάξει διεθνώς εντελώς το σκηνικό. Οι επενδύσεις στην ναυτιλία είναι αυξημένου ρίσκου, θέλουν ελάχιστες εγγυήσεις Γι' αυτό όπως ένας εφοπλιστής από τη δεκαετία του 1980 μου έλεγε όλοι τους θέλουν μια νομπρέλα για τις δύσκολες ώρες αλλά και για τις καλές ημέρες. Πρέπει κύριε Υπουργέ με την ευκαιρία αυτή να εντάχει ένας γρήγορος απολογισμός σε βασικούς τομείς κρίκους. Δηλαδή από το 1986 μέχρι τώρα η ναυτιλία σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολλαπλασιαστικά αυξήθηκε σε αριθμό πλοίων, σε μεταφορικό όγκο. Από την άλλη μεριά θα βρούμε ότι όλο και περισσότερο με πολύ γρήγορους ρυθμούς αντικαθίσταται το ναυτεργατικό δυναμικό με, φτηνότερο εργαζόμενο, με φτηνότερους εργαζόμενους. Τρίτος τομέας, βασικές ανάγκες των εσωτερικών μεταφορών και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την αυτοπλοεία της χώρας μας, μέχρι το 2002, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, δαπανούσε το ελληνικό κράτος 12 εκατομμύρια ευρώ. Και φτάσαμε πέρσι το 2013 να δαπανίσουμε για τις επιδοτήσεις των εφοπλιστών για τις άγωνες γραμμές 125 εκατομμύρια ευρώ. Άρα κάτι πηγαίνει στραβά εδώ. Και τέλος, να τελειώσω κύριε Πρόεδρε με το εξή. Είναι ανοιχτό το ζήτημα σε ό,τι αφορά με την απελευθέρωση των λιμενικών υπηρεσιών και το ξεπούλημα των λιμάνιων. Είμαστε ριζικά αντίθετοι. Θα πολεμήσουμε αυτή την εξέλιξη με όλες μας τις δυνάμεις, φυσικά με όρους κινήματος, ε, με τους πολιτικούς στο Ευρωκοινοβούλιο και στο Εθνικό Κοινοβούλιο. Κυρία Γκουλμάια, ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ε, θα σας καλωσορίζω και τους δύο. Φαντάζομαι είστε δύο γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλιά σας και βεβαίως είναι σαφές ότι κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας δίνετε μεγάλη έμφαση στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Αλλά καθώς ε, είμαι και σκιώδης ε, για ζητήματα της οίκων, ένα ερώτημα. Αναφερθήκατε λοιπόν ε, στη συμφωνία με το Συμβούλιο για ε, την ανάπτυξη ενός ε, διαπιχειρησιακού ευρωπαϊκού συστήματος. Μπορείτε να μας δώσετε περαιτέρω πληροφορίες για αυτό το σύστημα και ποια είναι τα ηχέγγυα για την αποτελεσματική και ομαλή λειτουργία ενός τόσο περίπλοκου ε, δικτύου. Θεωρώ ότι είναι ένα απαραίτητο τμήμα ε, για να μειωθούν ε, και τα ατυχήματα και ατυχή συμβάντα. Θα ήθελα να, να λάβω κάποιες απαντήσεις παρακαλώ και βεβαίως για την ελληνική προεδρία. Ο Πρωθυπουργό την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια έκανε μια εξαιρετική ομιλία και θέλω να πω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικά τόσο κάνατε γιατί έχετε, έχουμε τόσο υψηλή ανεργία στην Ευρώπη. Επομένως, ε, ελπίζω και εσείς να τα πάτε πολύ καλά, παρότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Γιάννα Σάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον Υπουργό για τις ε, πληροφορίες. Πρώτα απ' όλα, παρότι τέσσερις μήνες έχετε για μας ε, στην Προεδρία σας, Σημασία έχει η πολιτική βούληση. Διαρωτώ με κατά πόσο μπορείτε να μας δώσετε μια επισκόπηση της χρηματοδότησης των λιμένων στην Ευρώπη. Γιατί καθώς όπως έχουν φανεί από κάποια από αυτά τα ζητήματα, οι χώρες ε, και λιμένες ε, της Βόρειας Ευρώπης σε σχέση με τις Νότιας Ευρώπης ε, παρουσιάζουν πολύ σημαντικές διαφορές. Φαίνεται ότι ε, τα, οι της Νότιας Ευρώπης ε, πιέζονται και οδηγούνται ε, στο να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί. Δεν ξέρω αν υπάρχει επαρκής διαφάνεια. Ανησυχώ ότι δεν υπάρχει αρκετή διαφάνεια στον τρόπο χρηματοδότησης των λιμένων στο βορρά και στο νότο. Και αυτό θα διονύσει τις ανισότητες μεταξύ των δύο κατηγοριών. Θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική διαφορά μεταξύ Μεσογείου και Βαλτικής. Έτσι, μέχρι να υπάρξει πραγματική, πραγματικός ανταγωνισμός, ε, όσο υπάρχει ακόμα τόση φτώχεια και ανέχεια, είναι υπερβολικό. Ξέρω ότι σήμερα στην ε, Γερμανία υπάρχουν ε, κάποια ζητήματα όπως θέματα διαφθοράς. Βαθιά διαφθορά μαστίζει ολόκληρη τη χώρα. Επομένω θα ήθελα να σας ε, ρωτήσω. Αντί να δημιουργήσουμε λοιπόν αυτούς τους τεράστιους ε, υπερλιμένες με τελωνιακές ε, αρχές και από τρίτε χώρες, αν πρέπει να παρακολουθήσουν, να τηρήσουν μάλλον όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα, που είναι αυτό που μας ζητάει και η βιομηχανία, Αντί για αυτό λοιπόν, γιατί να μην ε, εξετάσουμε τα λεγόμενα clusters, κάποιους πυρήνες λιμένων που μπορούν να λειτουργήσουν από κοινού και έτσι θα μπορέσουν ε, να διεκπαιρεώσουν καλύτερους, πιο αποτελεσματικούς ε, και λιγότερο διαπανηρούς ελέγχους. Τέλος, τι, ε, ποια είναι η γνώμη σας για τις λεγόμενες λεωφόρους της θάλασσας και βεβαίως και για την διευκόλυνση συνδέοντας της στην Ευρώπη. Νομίζετε ότι αυτό μπορεί να επεκταθεί και στη Βόρεια Αφρική ή σε άλλες τρίτες χώρες. Και τέλος, για τα ναυπηγεία στην Ευρώπη, εσείς είστε χώρα ναυτική με μεγάλο εφοπλιστικό κλάδο. Θεωρείτε ότι μπορεί να, μπορούμε να δώσουμε ελπίδα στα ευρωπαϊκά ναυπηγεία. Και τέλος, ε, για την αλληλεία, ξέρω ότι ίσως σας, ε, να μην σας απασχολεί τόσο παρότι θα έπρεπε ως Έλληνες. Θεωρούμε ότι στην Ευρώπη θα έπρεπε να υπάρχει αλληλεία, να αυξηθούν οι ικανότητες και τα σκάφη. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζαβέλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώς ορίσατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλή επιτυχία στην ελληνική Προεδρία. Όπως γνωρίζετε, εδώ και δέκα μήνες περίπου, έχει αρχίσει η συνεργασία Ευρώπης-Αμερικής για την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Σίγουρα τα θέματα του εφοπλισμού, της ναυτιλίας και ιδιαίτερα θέματα που αφορούν το περιβάλλον, την αυτιλία, τα κρουαζερόπλια. Είναι θέματα τα οποία θα εξεταστούν στα πλαίσια αυτής της συμφωνίας. Προτίθεστε, έχετε καθόλου ενημερωθεί αν θα λάβετε μέρος σε κάποια από τις ε, συναντήσεις που συζητιέται αυτό το σύμφωνο ελευθέρου εμπορίου ε, της Ευρωατλαντικής Συμμαχίας. Ευχαριστώ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευρύ φάσμα ερωτήσεων κύριε Υπουργέ. Αν θέλετε να προσπαθήσετε τουλάχιστον να απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους βουλευτές που πήραν το λόγο και να πω σε όλους και σε καθένα ξεχωριστά που μου ευχήθηκαν ε, καλή επιτυχία. Ε, να, να σου ευχαριστήσω. Κοιτάξτε, είπαμε Προεδρία τεσσάρων μηνών, αλλά δεν είναι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Είναι έξι μηνών η Προεδρία. Το Κοινοβούλιο μόνο θα μας έχει εδώ για τέσσερις μήνες. Επομένως δεν είναι πραγματικά μια σύντομη Προεδρία. Είναι μια κανονική Προεδρία. Ε, σχετικά με τις ερωτήσεις και τα ζητήματα που, στα οποία αναφέρονται, γνωρίζω ότι υπάρχουν ήδη κάποια επίμαχα ζητήματα. Τα θέμα της απελευθέρωσης των λιμένων, αυτός ο κανονισμός, ο φίλος μου ο Γιώργος ε, το ονόμασε τον κανονισμό προβληματικό, δηλαδή ότι είχε προβληματικό παρελθόν. Είναι σαφές αυτό και με ρώτησε πού βασίζουμε, πού στηρίζουμε την φιλοδοξία μας, την αισιοδοξία. Ε, η κυρία Γιάλα Σέντερ ε, ρώτησε πολλά πράγματα σχετικά με το πώς θα πρέπει να προχωρήσει και το γιατί θα πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία. Στους τριμερείς διαλόγους ευελπιστούμε ε, ότι μπορεί να εξευρεθεί κοινό τόπος και μέσω διαλόγου είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι μπορούμε να βρούμε αυτόν τον κοινό τόπο. Είναι γεγονό ότι ο κανονισμό έχει προβληματικό παρελθόν. Είναι γεγονό επίση ότι υπάρχουν διαφορέ ανάμεσα στου λιμένες του Βορρά και στου λιμένες του Νότου. Είναι γεγονό επίση ότι ε, στην ε, ε, Μεσόγειο υπάρχουν ανταγωνιστικοί λιμένε σε τρίτε χώρε εκτό τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Ε, ε, ε, από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι μπορούμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Πρέπει να είμαστε φυσικά πολύ προσεκτικοί και σαν Έλληνας και όχι μόνο σαν Προεδρεύων σας λέω ότι είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αλλά ως Προεδρεύων πρέπει να σας πω ότι θα δουλέψουμε και ευελπιστούμε ότι τα, τα αποτελέσματα, η έκβαση του τριμερούς διαλόγου θα είναι σωστά. αναφερθήκατε στη θαλάσσια ανάπτυξη. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Αναφέρθηκε από πολλούς συναδέλφους ε, και από την κυρία Μάισερ και από τον κύριο Τούσα. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό να κατανοήσει κανείς ότι η Επίτροπος κυρία Δαμανάκη έχει κάνει πάρα πολλή δουλειά έτσι ώστε ε, να ε, ε, να συγκεράσει κατά κάποιο τρόπο όλη την υφιστάμενη νομοθεσία τις οδηγίες τις σχετικές και οπωσδήποτε εμείς θα δουλέψουμε σε στενή συνεργασία με την Επίτροπο την κυρία Δαμανάκη Οπωσδήποτε όμως θα δουλέψουμε και για το συγκεκριμένο σχεδιασμό έτσι όπως προκύπτει από την δικιά μας συζήτηση. και θα δούμε κατά πόσο θα, πρέπει, κατά πόσο θα προκύψει ανάγκη για ε, πανευρωπαϊκό ή περιφερειακό σχεδιασμό ή πώς θα μπορέσουν να συγκεραστούν τα δύο στοιχεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε, να δουλέψουμε μαζί έτσι ώστε να προωθήσουμε την πρόταση. Η γαλάζια ανάπτυξη οπωσδήποτε σχετίζεται και προκύπτει μάλιστα από την διακήρυξη της Λεμεσού και θα προσπαθήσουμε να επιτύχουμε συμπεράσματα Συμβουλίου τον Ιούνιο, καθώς επίσης και συγκεκριμένο χρονικό σχεδιασμό όσον αφορά το θέμα αυτά. Εκπομπές και ε, καθαρή ενέργεια για τις ε, μεταφορές. Δεν ασχολείται το δικό μου υπουργείο με τα ζητήματα αυτά. Ε, είναι το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών. Συμφωνώ πάντως με τον κύριο Κράμερ ότι το ζήτημα είναι σημαντικό. Υπάρχουν ε, θέματα εκπομπών, ε, ε, κυρίως όσον αφορά την κατανάλωση και την πόντιση υγρών αποβλήτων σε λιμάνια. Είναι σίγουρο ότι θέλουμε καθαρές μεταφορές και να σας πω ότι οι θαλάσσιες μεταφορές είναι πολύ καθαρότερες από τις χερσαίες μεταφορές ε, ακόμα και από τις μεταφορές ε, επισταθερών τροχιών, σιδηρο, σιδηροδρομικές μεταφορές κτλ. Με τις θαλάσσιες μεταφορές ε, οι συνολικές εκπομπές ε, για μεταφορά ίσου φορτίου είναι πολύ μικρότερες στις θαλάσσιες μεταφορές. Το Συμβούλιο θέλει οπωσδήποτε να υπάρξει ε, επιμήκυνση της οδηγίας για την καθαρή ενέργεια μέχρι το 2030. Γνωρίζω ότι υπάρχουν φωνές στο Κοινοβούλιο που επιμένουν στον χρονικό στόχο του 2020 και εδώ πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε κάποιο κοινό τόπο. Όσον αφορά την ε, φορολόγηση, το κατά πόσον πληρώνουν οι εφοπλιστές ε, ή δεν πληρώνουν, ο φίλος μου ο Γιώργος Σωτούσας το ανέφερε αυτό. Κοιτάξτε, η εφοπλιστική βιομηχανία ε, είναι, ξέρετε, μια ιδιάζουσα, έχει παρουσιάσει μια ιδιάζουσα κατάσταση όσον αφορά την φορολογία. Είναι tax free κατά κάποιο τρόπο ε, γιατί μπορούν να μετακινηθούν από την μία χώρα στην άλλη. Ξέρουμε επίσης ε, ότι σε πολλές περιπτώσεις που κυβερνήσεις προσπάθησαν να επιβάλλουν συγκεκριμένη φορολογία έφυγαν πολλές ναυτιλιακές ε, επιχειρήσεις και πήγαν σε άλλες χώρες. Εν πάση περιπτώσει αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια επενδύσεις και πρέπει ε, να συνεχίσουν έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται περισσότερους ε, μεταφορείς ε, με ευρωπαϊκή σημαία, να έχουμε όσο γίνεται περισσότερες ναυτιλιακές υπηρεσίες που θα είναι πραγματικά ευρωπαϊκές. Το ζήτημα της βιομηχανίας της κρουαζιέρας. ιδιαίτερα στην περιοχή της Μεσογείου αναπτύσσεται με τους ρυθμούς και ε, προσπαθούμε να βελτιώσουμε τις συνθήκες, να βελτιώσουμε την ε, χρήση των ακτογραμμών μας με ταυτόχρονη προσπάθεια διατήρησης του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ακριβώς λέμε ότι θα πρέπει ε, να δούμε και την πλευρά του τουρισμού. Του τουρισμού το θέμα της μετανάστευσης, ξέρετε, ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς αρμοδιότητα της δικιάς σας Επιτροπής, ωστόσο είναι αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου. Έχουμε την πρόταση για τον ε, καθορισμό των ε, αρχών ε, όσον αφορά την προστασία των εξωτερικών συνόρων, συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα με σκοπό την, θαλάσσια, την προστασία των θαλασσίων συνόρων. Αναφέρομαι εδώ βέβαια στο έργο της Frontex. Είναι ένα ενωσιακό ζήτημα. Ε, πρέπει να σας πω ότι εγώ είμαι και επικεφαλής ε, των ε, λιμενοφυλάκων, της ελληνικής λιμενοφυλακής και κατά αυτήν την έννοια Έχω, πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο κύριους ε, στόχους. Ε, η ακτοφυλακή ε, προστατεύει τα σύνορα αλλά ελέγχει κατά κάποιο τρόπο και τις κινήσεις στην θάλασσα. Γνωρίζετε ίσως ότι ο πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς έχει αναλάβει την πρωτοβουλία να δημιουργηθεί μια task force για την Μεσόγειο ε, και συζητήθηκαν οι κατευθυντήρες γραμμές ε, ήδη πέρσι στο Συμβούλιο μαζί με μια άλλη επιχείρηση ε, που θα αφορά την επιτήρηση των ακτογραμμών όσον αφορά μετανάστες που προσπαθούν να βρουν καλύτερες συνθήκες ζωής και τους οποίους όμως βοηθούμε ενδεχομένως να βρουν τις συνθήκες αυτές επανερχόμενοι στην πατρίδα τους. Τα μηνύματα πρέπει να είναι σαφή. Πρώτον, σώζουμε τις ζωές τους στις θάλασσες, αλλά εντωμεταξύ δεν μπορούμε και να ανοίξουμε διάπλατα τα σύνορά μας και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία προσπάθεια έτσι ώστε να δημιουργηθεί ε, ένα pull-over effect. About shipyards, I'm not... Όσον αφορά τα ναυπηγεία, οφείλω να σας πω ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου. Νομίζω ότι ε, είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, ε, αν δεν, λαμβάν, αν δεν ε, σφάλω. Επίσης όσον αφορά τις, τα ατυχήματα θα απαντήσει ο αρμόδιος. Επίσης ε, για τα θέματα της αλληλείας ε, δεν είναι, δεν είναι δικά μου αρμοδιότητα του Υπουργείου μου. Τώρα τα τρία στοιχεία τα οποία στα οποία αναφέρθηκε η κυρία Τζαβέλα ε, η συμφωνία με τις ΗΠΑ είναι πάρα πολύ σημαντική. Αναθεωρούμε τα συγγνώμη, ελέγχομαι τα αποτελέσματα των ε, συζητήσεων και της προόδου της ε, Κομισιόν, αλλά μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι δεν έχουν προκύψει συγκεκριμένα ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ναυτιλία, γιατί ε, αυτά τα ζητήματα ρυθμίζονται από την Συμφωνία Ανοιχτής Θάλασσας. Δεν ξέρω εάν λησμόνησα να απαντήσω σε κάτι συγκεκριμένο. Ε, προσπάθησα να σημειώσω όλα τα στοιχεία. Α, ναι, ε, το όρομα για την ε, Μεσόγειο. Το τελευταίο σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω. Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε μία ανοιχτή, ασφαλή, καθαρή Μεσόγειο που θα ανοίξει διάβλατα τις πόρτες της στον τουρισμό και που ταυτόχρονα θα είναι και μία θάλασσα ανάπτυξης. Γι' αυτό ακριβώς προωθούμε την ιδέα των θαλασσίων λεωφόρων έτσι ώστε να διασυνδεθούν όχι μονάχα οι λιμένες της Μεσογείου οι ενωσιακοί αλλά και οι μη ενωσιακοί να ξεπεραστούν όλα τα, τα ε, διοικητικά γραφειοκρατικά προσκόμματα ε, και βεβαίως ε, και το ζήτημα της γαλάζιας ζώνης φυσικά και αυτό εντάσσεται στην εικόνα, στην ιδέα, το όραμα που έχουμε για την Μεσόγειο. Ευχαριστώ κύριε Μάσινερ, αλλά σύντομα γιατί περιμένουμε και άλλο κόσμο και άλλον υπουργό. Ναι, ναι. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την στρατηγική για την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών. Εσύ είστε αρμόδιο, δεν μου δώσατε όμω απάντηση. Απάντηση. Ναι, έχουμε τον Υπουργό των Εξωτερικών που ασχολείται με το θέμα αυτό. Κύριε Βαρβιτσιώτη, κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, για τις απαντήσεις, ερωτήσεις των βουλευτών. Στη διάρκεια ολόκληρης λοιπόν της ελληνικής προεδρίας, έστω και αν είναι μόνο τέσσερις μήνες, σας περιμένουμε να τα ξαναπούμε. Πρόεδρος θα είστε ολόκληρη τη διάρκεια της θητείας. Σας ευχαριστώ θερμά λοιπόν που ήρθατε και για την ομιλία σας. Okay. Next colleagues, Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα έχουμε τον Υπουργό Μιχάλη Χρυσοχοίδη Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. απόφυτο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκη. Είναι τόσο επιστημονικό αυτό το όνομα του Πανεπιστημίου. Πάντα με εντυπωσίαζε. Εκλέγεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 1989. Κύριε Υπουργέ, ξέρω ότι ήσασταν πριν πρόεδρος ναυτιλίας, τώρα έχετε όλα τα στεγνά ήδη των μεταφορών. Και έτσι σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ. Thank you very much, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, Ευρωβουλευτές, είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ ενώπιόν σας για να παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας στον τομέα της αρμοδιότητάς μου που είναι οι υποδομές και οι μεταφορές. Θα ήθελα καταρχήν πριν παρουσιάσω τις προτεραιότητες μας να ευχαριστήσω θερμά ε, άλλες δύο χώρες, την Ιρλανδία και την Λιθουανία που μαζί με την Ελλάδα αποτέλεσαν το λεγόμενο τρίο της Προεδρίας και δούλεψαν για, για μια κοινή προγραμματική στόχευση. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τη Γραμματεία του Συμβουλίου αλλά και τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα για την υποστήριξη που είχαμε στο στάδιο της προετοιμασίας της ελληνικής προεδρίας. Ελπίζω και εύχομαι να έχουμε μια πρόσκοπτη συνεργασία για ένα δημιουργικό και παραγωγικό εξάμεινο. Η ελληνική προεδρία, όπως ξέρετε, έχει την ιδιαιτερότητα ότι είναι πολύ ε, μικρή σε διάστημα χρονικό λόγω των ευρωεκλογών αλλά ταυτόχρονα πολύ σημαντικά τα θέματα τα οποία καλούμαστε να διαπραγματευτούμε. Θα περάσω λοιπόν απευθεία στην ε, παρουσίαση των προτεραιοτήτων μου της Προεδρίας μας, ειδικότερα στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών. Η Ελληνική Προεδρία θα συνεχίσει με το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο, που επί της ουσίας αποτελεί μια νομοθετική δέσμη και ένα μέσον για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρομικού τομέα έναντι άλλων τρόπων μεταφοράς στην Ευρώπη. Αποτελεί εξάλλου δέσμευση της ελληνικής προεδρίας να χειριστεί το τέταρτο σιδηροδρομικό πακέτο ως μια πάρα πολύ σημαντική προτεραιότητα στον τομέα των χερσαίων μεταφορών. Στην κατεύθυνση αυτή θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στον τεχνικό πυλώνα της τέταρτης δέσμης για μέτρα για τους σιδηροδρόμους και πιο συγκεκριμένα στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού με αριθμό 881 του 2004. Είναι απόφασή μας να δουλέψουμε σκληρά για την πρόταση αυτή προκειμένου να επιτευχθεί μια γενική προσέγγιση στο Συμβούλιο Μεταφορών Τηλεπικοινωνιών και Ενέργειας το Μάρτιο του 2014 να επιτύχουμε μια πολιτική συμφωνία ανάλογα με το αν το Ευρωκοινοβούλιο γνωμοδοτήσει πριν από την ημερομηνία αυτή. Έτσι θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις εργασίες στο πλαίσιο του Συμβουλίου σχετικά με τον τεχνικό πυλώνα. Μετά το Συμβούλιο του Μαρτίου, πρόθεση της Ελληνικής Προεδρίας είναι να ξεκινήσουν σχετικά με το σκέλος του ανοίγματο της αγοράς του τετάρτου σιδηροδρομικού πακέτου, ενδεχομένως και μέσω της διοργάνωσης μιας πολιτικής συζήτησης. Το σημερινό μας πρόγραμμα προβλέπει έναξη των συζητήσεων σε επίπεδο Συμβουλίου με τις υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, όμως είμαστε σε συνεχή επαφή με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και καθώς η δυναμική μεταβάλλεται δεν αποκλείεται να αλλάξουμε και τη σειρά των φακέλων αν χρειαστεί. Σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμά μας είναι να παρουσιάσουμε αναφορά προόδου στο Συμβούλιο Υπουργών της 5ης Ιουνίου του 2014. Η αφοσίωσή μας στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών φαίνεται άλλωστε και από το γεγονός της ένταξης της προτεραιότητές μας και της πρότασης για, τη δημιουργία του Shift Rail. Του Shift to Rail. Πρόκειται για ένα θέμα εξαιρετικής σημασίας. Αφού αφορά άμεσα την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία, όλο τον τομέα των σιδηροδρόμων και φυσικά τον κόσμο της έρευνας στην Ευρώπη. Αν και το θέμα αυτό θα παρουσιαστεί στην Ήτρε, την άλλη επιτροπή, στόχος μας είναι να ολοκληρώσουμε τις εργασίες σε επίπεδο Συμβουλίου στις 14 Μαρτίου του 2014. Λόγω της νομικής μορφής της πρότασης, πρόκειται δηλαδή για πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου, απαιτείται η θετική γνώμη του Κοινοβουλίου. Εμείς θα συνεργαστούμε στενά με όλες τις πλευρές ώστε να εξασφαλίσουμε ότι όλοι μαζί βαδίζουμε προς την ίδια θεώρηση. Συνεχίζω τις προτεραιότητες της Προεδρίας με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Πρόκειται για ένα φάκελο μεγάλη σημασία αφού για πρώτη φορά έχουμε νομοθετική πρόταση για το σημαντικότερο θέμα της απεξάρτησης του τομέα μεταφορών από το πετρέλαιο μέσα από τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Άλλωστε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του στις 22 Μαΐου του 2013 συγκαταλέγει την έγκριση της οδηγίας αυτής μεταξύ των δράσεων προτεραιότητας που πρέπει να ληφθούν για τη διευκόλυνση των επενδύσεων και για την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η δημιουργία κατάλληλης υποδομής ανεφοδιασμού είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσουμε να, να, να ξεκλειδώσουμε τις δυνάμεις της αγοράς. Να δοθεί όθηση στη σχετική οικονομική δραστηριότητα, να δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά και να μειωθεί σημαντικά με αποδείξεις και με αριθμούς η εξάρτηση της Ευρώπης τόσο πολύ από το πετρέλαιο. Στην Λιθουανική Προεδρία έγινε μια σημαντική δουλειά στο φάκελο αυτό. Επετεύχθη κοινή προσέγγιση σε επίπεδο Συμβουλίου. Έγινε ο πρώτος τρίλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ελληνική προεδρία συνεχίζει εντατικά τις διαπραγματεύσεις με το Κοινοβούλιο στη βάση ενός σχεδίου επαφών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής, της Ελληνικής Προεδρίας με στόχο την ολοκλήρωση του φακέλου στις 5 Μαρτίου του 2014. Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά και θα μπορούμε στις 14 Μαρτίου στο Συμβούλιο να ανακοινώσουμε θετικά αποτελέσματα. Αναφορικά με τις αεροπορικές μεταφορές, συνεχίζουμε τις εργασίες για το αεροπορικό πακέτο. Αναγνωρίζουμε τη σημασία του νομοθετικού αυτού εργαλείου ως μέσο για την αντιμετώπιση των δύο μεγαλύτερων προκλήσεων των ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Της χωρητικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών και θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική την πρωτοβουλία και τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σπάσιμο του ευρωπαϊκού πακέτου, καθώς και την ταχύτατη και θεσμική ανταπόκριση του Συμβουλίου στην προτροπή του Κοινοβουλίου να αρχίσουν διαπραγματεύσεις για μια πρόταση στο θέμα του θορύβου. Η ελληνική Προεδρία, με αίσθημα ευθύνης, συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωκοινοβούλιο σε επικοδομητικό πνεύμα για την επίτευξη μιας συμφωνίας στο θέμα της πρότασης για το θόρυβο το συντομότερο δυνατόν και με τη βοήθεια όλων των εμπλεκομένων μερών. Στις προτεραιότητες μας επίσης για το θέμα των επιβατικών μεταφορών, των αεροπορικών επιβατικών μεταφορών, εντάσσουμε και τα δικαιώματα επιβατών με την πρόταση κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού 261 του 4 για τη θέσπιση κοινών κανόνων αποζημίωσης των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και παροχής βοήθειας σε αυτούς σε περίπτωση άρνηση επιβίβασης, ματέωσης ή μεγάλης καθυστέρησης πτήσης, καθώς και του κανονισμού 2027 το 97 για την ευθύνη του αερομεταφορέα όσον αφορά την αεροπορική μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους. Είναι κοινό τόπος πως οι ισχύοντες κανόνες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών πρέπει να αναθεωρηθούν, να αποκατασταθεί ένα πνεύμα δικαίου, να διασφαλιστεί η δίκαιη κατανομή βαρών και να επιτευχθεί τελικά η αποτελεσματική και μόνιμη εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων. Με πλήρη επίγνωση αυτού του φακέλου η Ελληνική Προεδρία προτίθεται να συνεχίσει την καλή δουλειά που ξεκίνησε από την προηγούμενη Λιθουανική Προεδρία και να φτάσει σε μια γενική προσέγγιση δεδομένου ότι παραμένουν ακόμη αρκετά εκρεμή ζητήματα. Επισημένω δε ότι δεδομένη της πολυπλοκότητας της πρότασης και το εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα πριν από το τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περίοδου δεν μπορούμε να θεωρούμε ρεαλιστικό στόχο την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων σε πρώτη ανάγνωση από τα δύο νομοθετικά όργανα, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόταση αυτή. Επίσης, στις προτεραιότητάς μας έχουμε εντάξει και την πρόταση οδηγίας για τα βάρη και τις διαστάσεις. Γνωρίζοντας πολύ καλά πως πρόκειται για μια πρόταση της Επιτροπής με αμφιλεγόμενα στοιχεία. Παρ' όλα αυτά η Προεδρία μας προτίθεται να εργαστεί εντατικά και επικοδομητικά με σκοπό την επίτευξη γενικής προσέγγισης μέχρι τον Ιούνιο του 2014. Παρά το γεγονός ότι εμείς ως χώρα δεν διαθέτουμε πλωτούς ποταμούς. Είμαστε μια ναυτική χώρα. Η Προεδρία μας θα ασχοληθεί με την πρόταση κανονισμού για την τροποποίηση του κανονισμού 718 του 1999 για την πολιτική και τη χωρητικότητα του κοινοτικού στόλου για την προώθηση των εσωτερικών πλωτών μεταφορών. Η πρόταση είναι κατατέθη ως τμήμα της συνολικής πρότασης Ναϊάδες το φθινόπωρο του 2013. Σεβόμενοι απολύτως το γεγονός ότι αυτές οι μεταφορές έχουν τεράστια αναπτυξιακή σημασία για πολλές χώρες της Ένωσης, αποφασίσαμε να συζητήσουμε την πρόταση στο Συμβούλιο με στόχο την επίτευξη κοινή προσέγγισης στο Συμβούλιο της 5ης Ιουνίου το 2014. Τέλος, ανάλογα με την πορεία των εργασιών και τις σχετικές διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη, η Προεδρία θα διερευνήσει και τη δυνατότητα για επεξεργασία και έγκριση συμπερασμάτων για την ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την αστική κινητικότητα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη φυσικά και τους χρονικούς περιορισμούς που έχει η τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδος λόγω των εκλογών. Ωστόσο, ζητούμε τη δική σας συνδρομή, τη δική σας συνεργασία, τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων μερών και θεσμών και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ θετικά ε, αποτελέσματα για τους κέριους τομείς της πολιτικής μεταφορών που αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες για την ανάπτυξη στην Ευρώπη που είναι το ζητούμενο της εποχής μας μιας και μέσα από την ανάπτυξη θα καταπολεμήσουμε τα κοινωνικά προβλήματα μα κυρίως την ανεργία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα μόνο να αναφέρω τους ομιλητές Γκρός, Αλκαντράουι, Μάισνερ, Κράμερ, Μπακ, Σαναλόβα, Μπιλμπάο, Δανέλης, Αγιάλα, κύριος Κουμουτσάκος. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο να προσταθεί στον κατάλογο, την Τάντζα. Εντάξει. Προτείνω να θέσουμε τέσσερα λεπτά για τους συντονιστές και μετά δύο λεπτά για τους υπόλοιπους ομιλητές. Ο κύριος Γκρός πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και ευχαριστώ κύριε Προεδρεύον. Σας ευχαριστώ πολύ για τις δηλώσεις και τις παρατηρήσεις σας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και ιδιαίτερα στις διαπραγματεύσεις. Έχετε φτάσει να διαπραγματεύεστε πέντε συμφωνίες και μια έκθεση προόδου σε διάφορα θέματα που θα έλεγα είναι επιδόσεις ολυμπιακές. Άθλος μεγάλος που θα πρέπει να επιτελέσετε μέσα στους τέσσερις μήνες. Πάντως να ξέρετε πάντα ότι είμαστε στο πλευρό σας και η Επιτροπή σας στα πολύ σημαντικά αυτά θέματα που έχουν σημασία όχι μόνο για τις μεταφορές αλλά και για την οικονομική ανάπτυξη και άλλα σημαντικά ζητήματα ε, ιδιαίτερα για ορισμένα κράτη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είμαστε στρατευμένοι στην προώθηση των θεμάτων αυτών και ιδιαιτέρως μας ενδιαφέρει να μην καθυστερούν τα ζητήματα αυτά και τα έργα αυτά στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο έχει καλές προτάσεις και πιστεύω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε με αυτές σε καλές συμβαστικές λύσεις για να καταλήξουμε σε τελικές συμφωνίες, final agreements. Ε, είναι καλά τα θέματα, είναι ενδιαφέροντα τα θέματα. η πτυχή του περιβάλλοντος αλλά και η πτυχή της ασφάλειας στα οχήματα πρέπει να τεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων. Και βεβαίω έχουμε όλο, όλη τη δέσμη των προτάσεων για τα σιδηροδρομικά, για το σιδηρόδρομο. Είναι το πακέτο το σιδηροδρομικό ιδιαίτερη προτεραιότητα, όπω μα είπατε. Και εμεί είμαστε πεπισμένοι ότι ο σιδηρόδρομο δεν θα είναι απλώ μια καλή εναλλακτική για την Ευρώπη, μαζί βέβαια με τι θαλάσσιε μεταφορέ, αλλά ιδιαίτερα ε, μπορεί να έχει ένα τεράστιο δυναμικό απασχόληση. Εάν αναπτυχθεί ο σιδηρόδρομο, μπορεί να βοηθήσει ιδιαίτερα στην αύξηση των θέσεων απασχόληση. Και πολύ σωστά ε, πρέπει να ξεκινήσει κανείς από το τεχνικό πεδίο. Αλλά μην ξεχνάμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια δέσμη, ένα σύνολο προτάσεων. Ξέρουμε ποιο είναι ο κύριο κίνδυνο, ο μεγάλο κίνδυνο να κατακαιρματιστεί το πακέτο αυτό, διότι έχει μια ε, παράξενη τάση το Συμβούλιο να διαλέγει τα κομμάτια που του αρέσουν και τα άλλα να τα αφήνει για τις ελληνικές καλένδες. Παρακαλώ λοιπόν πείτε στο Συμβούλιο ότι πρέπει να προχωρήσει κατά προτεραιότητα και το πακέτο αυτό ε, πολύ γρήγορα για να ολοκληρωθεί όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Ο συνάδελφος Μπαχ έχει ασχοληθεί με το θέμα των δικαιωμάτων των πολιτών, των επιβατών συγκεκριμένα. Ο εισηγητής είναι κάτι το οποίο όπως γνωρίζετε μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Εγώ τώρα έχω μια ερώτηση σχέση με τις αεροπορικές μεταφορές, όπου πάλι μια και το θέμα της ηχορύπανσης του θορύβου ε, το αναφέρατε και εσείς, αλλά νομίζω ίσως όχι τόσο όσο στα άλλα μέσα, θα ήθελα να ρωτήσω για το θέμα των σλότς, των χρονοφυρίδων. Είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να προχωρήσει από ένα πρώτο τριμερή διάλογο που είχαμε να προχωρήσουν τα θέματα της ηχορύπανσης και των χρονοθυρίδων. Ε, επίσης, έχουμε το μέσων ε, συνδέοντας την Ευρώπη, Connecting Europe Facility. Έχουμε την κυρία Αγιάλα, τον κύριο Κουμουτσάκο που έχουν ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα θέματα αυτά των ε, διευρωπαϊκών δικτύων που πρέπει να προωθηθούν και θα ήθελα να σας ρωτήσω τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Και μια τελευταία ερώτηση, ιδιαίτερα για μια χώρα όπως η Ελλάδα που έχει τεράστιες προκλήσεις μπροστά τη και οικονομικές βέβαια αλλά και σε επίπεδο υποδομών. Πώς το βλέπετε αυτό ως προεδρεύων το σύνολο και πώς μπορείτε εσείς να αξιοποιήσετε και να υλοποιήσετε τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αλκαντράου έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Υπουργό για την εισαγωγή του, να σας ευχαριστήσω και να σας ευχηθώ πολύ καλή επιτυχία για τους επόμενους μήνες. Η Προεδρία βεβαίω και θα διαρκέσει έξι μήνε, αλλά η περίοδο κατά την οποία θα υπάρξουν και διαπραγματεύσει με το Κοινοβούλιο είναι πραγματικά πολύ περιορισμένο. Θα επικεντρωθώ σε δύο θεματικές. Πρώτον για τους σιδηροδρόμους και δεύτερον αεροπορία. Αεροπορικές μεταφορές. Για τους σιδηροδρόμους ε, το θέσατε κι εσείς ως βασική προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας. Θα ήθελα να πω βέβαια ότι δεν φταίτε εσείς γι' αυτό, αλλά συνδέεται με τη λειτουργία του Συμβουλίου. Απογοητευθήκαμε από τις καθυστερήσεις κατά τις διαπραγματεύσεις στο ιστορικό του Συμβουλίου για το πακέτο αυτό. Εμείς καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια, κάναμε τα δύνατα δυνατά για να εργαστούμε σε αυτό το ευαίσθητο και εξαιρετικά εκτεταμένο πακέτο. Βεβαίως ακολουθούμε διαφορετική τεχνική. Πρώτα εξετάζουμε τα τεχνικά και μετά περνάμε στους πιο πολιτικούς ε, φακέλους. Αλλά ε, είχαμε ελπίσει πριν από το τέλος ε, της κοινοβουλευτικής μας τουλάχιστον να υπάρξουν διαπραγματεύσεις και να υπάρξει συμφωνία για το τεχνικό πακέτο. Μόλις το Συμβούλιο του Μαρτίου θα μπορούσε να γίνει ένας μια συζήτηση προσανατολισμού. Είναι πολύ αργά για να υπάρξει συμφωνία κρίμα. Εμείς ε, θέλαμε να μοιράσουμε κάπως αυτή τη συζήτηση. Πρώτα να ξεκινήσουμε με, τα, με τον τεχνικό, τους τεχνικούς δείκτες, αλλά δυστυχώς αυτός δεν θα γίνει. Αυτό δεν θα γίνει. Τώρα, για την ε, αεροπλοεία, μιλήσατε για το πακέτο των αεροδρομίων. Αυτό έχει ολοκληρωθεί εδώ και πολύ καιρό σε εμά. Δεν αφορά μόνο το θόρυβο, αλλά και κοινωνικούς ε, κανόνες ε, στις υπηρεσίες εδάφους και για το πώς θα αναγνωρίζονται στο, μέλλον ε, οι χρονοθερίδες. Εμείς είμαστε διαθετημένοι να διαπραγματευτούμε από αυτού ξεχωριστά γιατί ξέρουμε ότι για τα υπόλοιπα δεν είστε ακόμα έτοιμοι και δεν μπορείτε να, συνεχίσετε, να ξεκινήσετε τις συζητήσεις. Ελπίζουμε τουλάχιστον για το θόρυβο να μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόοδο. Για τα δικαιώματα των επιβατών ε, του συναδέλφου Μπαχ είναι αυτός ο φάκελος. Ε, τον επόμενο μήνα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια σε μερικές εβδομάδες και θα λάβουμε τελική οριστική θέση. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια μοναδική ευκαιρία να δείξουμε στον Ευρωπαίο πολίτη ότι η Ευρώπη με πολύ συγκεκριμένο τρόπο μπορεί να έχει απτά αποτελέσματα, να προστατεύσει τον πολίτη και σε περίπτωση προβλημάτων να μερευνήσουμε τόσο ώστε να έχουν την κατάλληλη ε, φροντίδα και στήριξη. Και θα σας καλούσα να κάνετε ό,τι μπορείτε για να ε, σημειωθεί ως τον μεγαλύτερη πρόοδος σε αυτόν τον φάκελο. Τελευταίος φάκελος ε, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών είναι ο τομέας του ενιαίου εναέριου χώρου. Βεβαίως εδώ και πολλά χρόνια μας απασχολεί αυτό το ζήτημα. Εμείς μόνο διαπιστώνουμε ότι η νομοθεσία που έχει ήδη εγκριθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το Single European Sky δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί στην πράξη παρότι μένουν πολλά ακόμα να γίνουν για το περιβάλλον αλλά και για τη βιομηχανία σε τη φορά την μείωση του κόστους και σε ό,τι αφορά την αποδοτικότητα, το οποίο βεβαίω ωφελεί και του επιβάτε. Τώρα, τουλάχιστον με αυτό το Single European Sky 2, μέχρι να εφαρμοστεί αυτό, για να εφαρμοστεί αυτό, θα θέλαμε και από εσά ε, να σημειωθεί μεγαλύτερη πρόοδο. Καλή επιτυχία λοιπόν, είμαστε στη διάθεσή σα να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστώ εκ μέρου των φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εγώ για την τοποθέτησή σας. Βεβαίως έχει σημειωθεί ότι η Προεδρία κρατάει έξι μήνες. Για μας οι τέσσερις είναι οι πρώτοι μήνες, μετά κλείνει το Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, στο θέμα των σιδηροδρόμων δεν θα τοποθετηθώ τώρα, γιατί συνάδελφος Μπιλμπάου Μπαραντίκα, ναι, εγώ είμαι η Μάισνερ, η κυρία Μπιλμπάου Μπαραντίκα θα μιλήσει στο θέμα αυτό, με το οποίο ασχολείται ιδιαίτερα ω συγγήτρια. Για τις υποδομές, θα ήθελα να πω δύο λόγια. Αναφέρατε τις υποδομές για εναλλακτικά καύσιμα. Εγώ έχω συμμετάσχει και στον τριμερό διάλογο, είμαι και σκιώδη συγγήτρια εκ μέρου τη ομάδα μου τη πολιτική και πιστεύω ότι θα ήταν ε, δυνατόν να εξασφαλίσουμε στις 5 Μαρτίου συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Έχουμε έτσι ένα καλό δείγμα και μια, ένα καλό μήνυμα και μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε περαιτέρω ώστε να εξασφαλίσουμε πιο υγιείς μεταφορές όπως το εννοεί και η Λευκή Βίβλος. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αναπτύξουμε αυτές τις υποδομές. Για τις ε, αεροπορικές μεταφορές πολλά ήδη υπόθηκαν, θα είμαι σύντομη. Ασφαλώς πρέπει να ξεκινήσουμε από το θέμα του ε, θορύβου, τη συγχωρήπανση, πάρα πολύ σημαντικό όπως το είπατε, αλλά και οι χρονοθυρίδες υπάρχει και εδώ ε, ανάγκη να προχωρήσουμε στο ενιαίους ευρωπαϊκούς εθέρες, Single European Sky. Θα συμφωνήσω με τον Σνάλφο Αλκαντράουι πρέπει να προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση στο θέμα αυτό και όπως και με τους σιδηροδρόμους χρειαζόμαστε λογικές λύσεις και για τις αεροπορικές μεταφορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπορείτε κάτι να επιτύχετε μέσα στην Προεδρία σας. Για τα δικαιώματα των επιβατών, όπου έχω ένα συγκεκριμένο ερώτημα. Δεν έχει κλείσει το θέμα βέβαια από πλευρά του Κοινοβουλίου ακόμα, δεν έχει ψηφιστεί, αλλά θέση του Κοινοβουλίου ε, που είναι πάντα πιο κοντά στον καταναλωτή από ό,τι η Επιτροπή. Ε, έχει οριστεί η περιπτώσει θέση του Κοινοβουλίου. Θέλω να ρωτήσω το Συμβούλιο πώ στάσατε στην υπόθεση αυτή. Και μια τελευταία ερώτηση. Εσεί είσαστε αρμόδιο υπουργό και για τον ΑΙΑΔΕ, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα την πολιτική μου ε, ομάδα και θα ήθελα να ακούσω λίγο πιο πολλά πράγματα. Ευχαριστώ ο κύριος Κράμερ και εγώ ευχαριστώ εκ μέρους της ομάδας των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ε, ομιλία σας, για τις ε, προτάσεις σας. Θα ήθελα ωστόσο να ακούσω και μερικά λόγια για την έκθεση Λίχτεμπερκ και τη δική μου για τις στατιστικές ε, στους σιδηροδρόμους και τις θαλάσσιες οδούς. Είναι κάτι το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ, δεν το βλέπω να προχωράει. Είναι στην ημερήσια διάταξη το επόμενο εξάμεινο. Επίσης χαίρομαι ιδιαίτερω που τοποθετηθήκατε για το πακέτο των σιδηροδρόμων. Είπατε ότι είναι κύρια προτεραιότητα για σας, διότι οι πληροφορίες που είχαμε από το περιβάλλον σας έδειχναν ότι η ελληνική προεδρία δεν ενδιαφέρεται για το θέμα αυτό και δεν πρόκειται να το προωθήσει. Άρα κατάλαβα καλά ότι για σας ο επόμενος πυλώνας είναι να προχωρήσει το τεχνικό κομμάτι, γιατί έχει καταλήξει το Συμβούλιο σε μία λύση για την διαλειτουργικότητα, interoperability και για την ασφάλεια, safety. Αυτά λοιπόν έχουν προχωρήσει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι προχωράνε γρήγορα και μπορούμε να πάμε στον τριμερή διάλογο για να κλείσουν αυτά τα θέματα και όπως είπε και ο Ματσιέ Γκρός να προχωρήσει ολοκληρωμένα το θέμα. Αλλά τουλάχιστον να ξεκινήσουμε έτσι γιατί έχει μόνο τέσσερις μήνες διάθεση το κοινοβούλιο. Βλέπω να γλέφετε καταφατικά. Αυτό πολύ με χαροποιεί. Μακάρι να το επιβεβαιώσετε. Γιατί και χθε μας απασχόλησε εδώ στην Επιτροπή και θα αποτελέσει φυσικά πολύ σημαντικό βήμα προόδου αν το καταφέρουμε. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολε διαπραγματεύσει, αλλά πρέπει να προχωρήσουν έστω και αν κοπεί σε κάποιο κομμάτι το, το, το κεφάλαιο, το τομέα αυτών των σιδηροδρόμων, θα ήθελα να προχωρήσει πολύ καλά σε όλα. Ευχαριστώ και περιμένω την απάντησή σα. Θα ήθελα οι, επόμενοι ομιλητέ να μιλήσουν μονάχα δύο λεπτά. Δύο λεπτά, ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, δώσατε μεγάλη σημασία στις ε, μεταφορές τις υπογραμμίσατε ιδιαίτερως. Νομίζω ότι είναι σοβαρό αυτό το καθήκον που αναλαμβάνετε, το χαρτοφυλάκιο. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Δυστυχώς τους τελευταίους μήνες και τα χρόνια το Συμβούλιο δεν είχε δώσει σημασία στα διάφορα θέματα των μεταφορών, αεροπορικές μεταφορές, σιδηροδρόμους, ένα αέριος ευρωπαϊκός χώρος. Δεν, αντιθέτως πάταγε φρένο συνέχεια το Συμβούλιο. Αυτό λοιπόν το οποίο μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, θίγει ήδη σε ένα βαθμό. Με χαρά ακούω ότι είναι πρώτη στην προτεραιότητα για σας. Είπατε ότι στις αρχές Ιουνίου ή μάλλον μέχρι τον Ιούνιο θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμφωνία. Ερωτώ λοιπόν και συνεχίσω από, από τα όσα ρώτησε η κυρία Μάισνερ, ποια είναι η δική σας θέση βλέπετε να τάσεστε πιο πολύ στο πλευρό της Κομισιόν, δηλαδή πιο πολύ υπέρ του κλάδου ε, του οικονομικού ή πιο πολύ υποστηρίζετε τα συμφέροντα των επιβατών όπως θα θέλαμε εμείς γιατί θα θέλαμε να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα προς τους ε, πολίτες και τους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει μια τοποθέτηση γενική από το Συμβούλιο η οποία θα είναι σαφής και υπέρ των επιβατών. Επίσης για τους σιδηροδρόμους είπατε ότι και εδώ δεν βλέπω καμιά ιδιαίτερη δυσκολία για τα τεχνικά θέματα. Είπατε ότι έχουμε ξεκινήσει τα τεχνικά θέματα. Ξέρω ότι είναι πολύ σημαντική βέβαια η σιδηροδρόμη και για, τον, για, το λεγόμενο κλάδο των σιδηροδρόμων, το, το industry. Ε, ωστόσο υπάρχει μια αμφισβήτηση ως προς τη σειρά που θα ακολουθηθεί, το PSO, τις ε, υπηρεσίες, ποιο απ' όλα θα εξεταστεί πρώτο. Γιατί μπορεί να αλλάξει η σειρά από ό,τι ακούγεται. Και από τι θα εξαρτηθεί η σειρά με την οποία θα συζητηθούν τα θέματα. Καταρχά, λοιπόν, ρωτώ εάν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Και δεύτερον, εάν όντω υπάρχει αυτή η σειρά και μπορεί να αλλάξει η σειρά, από τι θα εξαρτηθεί η αλλαγή σειρά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σεναλόβα. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, σε ευχαριστώ. Έχω μια ερώτηση από το χώρο των, ε, της ασφάλειας της μεταφορές. Άκουσα ε, τις ε, παρατηρήσεις για τις φιλοδοξίες ε, που έχετε σε περίπτωση αντιμετώπισης συνεπειών ε, τροχαίου ατυχήματο είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Ασφαλώ πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των δυστυχημάτων, τον αριθμό των νεκρών στου ευρωπαϊκού δρόμου. Ιδιαίτερα λοιπόν το e-call μπορεί να είναι μια προτεραιότητα, πρέπει να είναι μια προτεραιότητα και θα ήθελα ιδιαίτερα να σημειώσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να υποστηρίξει και το έχει ήδη δηλώσει σαφώ την εισαγωγή του e-call. Είχαμε από τον Ιούλιο του 2012 με μια έκθεση που εγκρίθηκε σημειώσει και μάλιστα εγώ την είχα αναλάβει μαζί με τον συναρφό Κόχο ότι πρέπει να ενταχθεί από τον Οκτώβριο του 2015 στο σύστημα, το σύστημα αυτό να εισαχθεί. Γιατί λοιπόν να καθυστερούμε. Κάθε καθυστέρηση κοστίζει ζωές ανθρώπινες για τις ε, υποδομές. Τα έργα 1 και 2 βεβαίως βλέπω ότι έχουν προχωρήσει καλά και αναλόγως με, τις, ε, με τη στάση που έχουν τηρήσει τα ε, επιμέρους κράτη. Πώς μπορούμε λοιπόν να δούμε την ε, συνεργασία για να ολοκληρωθεί σε πρώτη ανάγνωση το θέμα αυτό, σε συνεργασία λοιπόν με το Κοινοβούλιο. Δύο λεπτά η κυρία Μπιλμπάου, πάρα πολύ σύντομα. Πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον Προεδρεύοντα και να ευχηθώ τα καλύτερα για την Προεδρία. Με μεγάλη χαρά ακούσαμε ότι η τέταρτη δέσμη των σιδηροδρόμων εντάσσεται στα μιλήματα της ελληνικής Προεδρίας γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως είχαμε ακούσει διάφορες, διάφορες φήμες ότι δεν ενδιαφέρεται η ελληνική Προεδρία γι' αυτό. Αναβερθήκατε στο γεγονός ότι το Μάρτιο ίσως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τα τεχνικά ζητήματα. Κοιτάξτε, ε, έχει καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια από πολλούς ε, βουλευτές ε, και ε, φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει δυσκολία όσον αφορά αυτά τα ζητήματα. Πάντως το ε, Συμβούλιο κατάφερε κάτι που προσπαθούσε το Κοινοβούλιο να ε, αποφύγει, να κάνει δηλαδή το διαχωρισμό πολιτικών και τεχνικών ε, θεμάτων. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προχωρήσουμε οπωσδήποτε και το πολιτικό και αυτή η ημερομηνία του Ιουνίου δεν μας βολεύει γιατί δεν θα, θα έχουν σταματήσει οι εργασίες στο Κοινοβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, ε, ε, εσείς στο Συμβούλιο τι ακούτε από τα κράτη-μέλη βλέπετε να υπάρχει κάποια διάθεση πραγματικής προόδου ε, του, της δέσμης ε, για τους ε, σιδηροδρόμους από τα κράτη-μέλη και όσον αφορά πολιτικό σκέλος, ποιες είναι κατά την άποψή σας οι μεγαλύτερες δυσκολίες έτσι ώστε να μην μπορέσει να φτάσει το θέμα στο Κοινοβούλιο πριν από την ημερομηνία που είπατε. Κύριε Δανέλη, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Ε, Καλώς όρισατε αγαπητέ μου Υπουργέ. Θέλω να ευχηθώ στην Ελληνική Προεδρία να είναι ε, επικοδομητική και αποτελεσματική. Και σε πολύ μεγάλο βαθμό ε, η αποτελεσματικότητα θα εξαρτηθεί βεβαίως από την, ε, την πρόθεση των εκκρεμών ζητημάτων, την επίτευξη συμφωνιών μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και βεβαίως ορίμασης των ζητημάτων που θα λύσει η επόμενη Προεδρία. Ε, πρέπει να ήδη να αντιληφθήκατε ότι στην Επιτροπή μας σε πολύ μεγάλο βαθμό υπάρχει συνένεση, κοινή ε, αντίληψη ιεράρχηση των βασικών προβλημάτων και γι' αυτό να είστε βέβαιος ότι θα είμαστε επικοδομητικά στο πλάι της ελληνικής προεδρίας στο βαθμό που εκείνη θα προωθήσει τα ζητήματα ε, στα οποία αναφερθήκαμε. Θα κάνω δύο τηλεγραφικές αναφορές σε δύο ζητήματα, πολύ κρίσιμα νομίζω. Το πρώτο έχει να κάνει με τον ενίο ευρωπαϊκό ουρανό. Είναι αδιανόητο να συνεχίζουν τα κράτη-μέλη να θεωρούν ότι μπορούμε να, να διατηρούμε και να συντηρούμε 28 συν 10 ε, ε, συστήματα διαχείρισης ανέρειας πληροφορίας. Είναι αδιανόητο να αρνούνται πεισματικά κολλησιεργώντας τον απόλυτο εξορθολογισμό τον οποίο απαιτεί, απαιτούν οι εναέρειες μεταφορές. Ε, για λόγους εξοικονόμησης χρήματος, χρόνου και βεβαίως αντιμετώπισης προβλημάτων ε, περιβαλλοντικών η ελληνική προεδρία πρέπει να ξεκολλήσει αυτό το θέμα. Και να πω ότι στην Επιτροπή μας διαμορφώνεται η άποψη ότι θα μπορεί το, εξαιρετικά χρήσιμο αυτό πακέτο να προχωρήσει χωρίς το σκέλος των, των, της απελευθέρωσης των, των ε, ε, υποστηρικτικών υπηρεσιών. Ας αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία και να προωθήσετε ε, το ζήτημα αυτό παίρνοντας προσωπικά εσείς το θέμα στη διαχείρισή του να, να προσθέσω ότι η Ελλάδα είναι διανόητο ως χώρα ε, με, με εξαιρετική τουριστική βιομηχανία, της οποίας η βιομηχανία εξαρτάται κυρίως από τις αεροπορικές μεταφορές, να μην προωθεί τον εξορθολογισμό του ζήτηματος αυτού. Κλείνω λέγοντας ότι το πακέτο των δικαιωμάτων των επιβατών, παρότι είναι στο αρχικό στάδιο, είναι πολύ κρίσιμο να επισπευθεί, διότι στέλνει και ένα μήνυμα πολιτικό στον Ευρωπαίο πολίτη, ότι η Ένωση ασχολείται και με καθημερινά ζητήματα βελτίωσης των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν. Ευχαριστώ πολύ. Αγιάλα Σέντερ, δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλώς ορίσατε κύριε Υπουργέ και ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σχετικά ε, με την ε, κοινή επιχείρηση Shift to Rail. σε αυτήν την ε, πλατφόρμα. Την τελευταία στιγμή ε, υπήρξαν ε, δυσλειτουργίες. Υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις από κράτα μέλη και από τη χώρα μου αλλά και από την Πολωνία και από τη Γαλλία που ήθελαν να συμμετάσχουν. Πιστεύω ότι αυτή η πλατφόρμα η οποία θα έπρεπε να είναι η πιο ισχυρή, όσο γίνεται πιο δυνατή λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες ε, θα πρέπει να ε, έχουν σε αυτήν την πλατφόρμα τη δυνατότητα ε, ανταγωνιστικές εταιρείε να μπορούν να συμμετάσχουν. Επίσης, όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, προηγουμένως θα ήθελα να επανέλθω σε, αυτήν, σε αυτό το θέμα της interoperability και της, της διατροπικότητας αλλά και της ασφάλειας. Μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα ζητήματα αυτά και όπως είπαν και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, μας ενδιαφέρει πολύ στη δέσμη των σιδηροδρόμων να προχωρήσει ε, το πολιτικό σκέλος ε, ε, γνωρίζοντας το προφίλ σας, γνωρίζοντας την παρούσα κατάσταση, ίσως μπορείτε να μας δώσετε ε, και κάποιες ε, επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την διευκόλυνση Connecting Europe, συνδέοντας την Ευρώπη και εδώ θα πρέπει να ξεκινήσουν οι επαφές όσο γίνεται πιο γρήγορα όσον αφορά τις, τους διαδρόμους, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία, να ξεκολλήσει. Όσον αφορά τώρα τα δικαιώματα ε, των, επιβατών θα πρέπει να φτάσουμε στις εκλογές με κάποια καλά νέα. Νομίζω ότι ε, ξέρετε πόσο δύσκολη θα είναι η προεκλογική εκστρατεία και επομένως θα πρέπει να έχουμε κάποια χαρτιά στα χέρια μας. Νομίζω ότι το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο κύριος Κουμουτσάκος, δύο λεπτά. Γιώργο, έχεις δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Μεταφορών. Σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο και απαιτητικό έργο τη Προεδρία, δεδομένου ότι νομοθετικά το έργο σα και η αποστολή σα συμπιέζεται σε τέσσερι μήνε λόγω των ευρωπαϊκών εκλογών. Ε, η Επιτροπή αυτή, όπω τα έχετε ήδη αντιληφθεί, θα στηρίξει την προσπάθειά σα και με την τεχνογνωσία που διαθέτει, αλλά κυρίω με την πολιτική τη βούληση να δει πρόοδο σε πολύ σοβαρά θέματα για τι ευρωπαϊκέ μεταφορέ. Δύο θέματα θέλω να θίξω, ε, κύριε Υπουργέ. Ε, άκουσαμε ε, πολύ θετικά το γεγονός ότι έχετε βάλει ψηλά στην προτεραιότητά σας το θέμα της προόδου στο φάκελο Ναϊάδες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, για τις ε, διατροπικές συνδυασμένες μεταφορές σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό συνδέεται με το άλλο και δεύτερο και τελευταίο θέμα που θέλω να αναδείξω. Με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. κύριε Υπουργέ, έγινε μια μεγάλη δουλειά τα τελευταία χρόνια. Αποφασίστηκε το νομοθετικό πλαίσιο. Υπάρχει το χρηματοδοτικό εργαλείο Είμαστε τώρα στη φάση της εφαρμογής. Για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή αυτού του μεγάλου, ίσως του μεγαλύτερου αναπτυξιακού σχέδιου υποδομών της Ευρώπης για τα επόμενα 15 χρόνια, έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω ότι με την δυνατότητα του καθεστώτος της προεδρεύουσας χώρας θα πρέπει να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας για να ξεκινήσει το ταχύτερο αυτή η εφαρμογή. Με επαφέ με την Επιτροπή, με μια τεχνογνωσία που χρειάζονται τα κράτη-μέλη, κυρίω τα κράτη-μέλη συνοχή. Η Ελλάδα, λόγω και αναφέρομαι μόνο στη χώρα μου θα μου το επιτρέψετε, λόγω γεωπολιτική θέση έχει μια χρυσή ευκαιρία να γίνει ένα ευρωπαϊκό και διεθνή διαμετακομιστικός κόμβο. Αλλά δεν φτάνει η γεωπολιτική θέση, χρειάζεται και υποδομέ. Και τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και το χρηματοδοτικό εργαλείο συνδέοντα στην Ευρώπη τη δίνει μια μεγάλη δυνατότητα, είναι μια μεγάλη ευκαιρία και η εκκίνηση τη εφαρμογή αυτού του μεγάλου σχεδίου, αναπτυξιακού σχεδίου, είναι εξαιρετική σημασία και για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Φιντάντζα, δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θα ενώσω τη φωνή μου στην φωνή όλων όσων ευχήθηκαν στην ελληνική προεδρία καλή επιτυχία. Είναι φιλόδοξο το πρόγραμμα και βεβαίως για μας τους Ιταλούς είναι διπλά σημαντικό αυτό το πρόγραμμα γιατί θα πάρουμε τη σκητάλη από την ελληνική προεδρία και επομένως πραγματικά σας εύχομαι όσο γίνεται περισσότερα να καταφέρετε εσείς. Καλή επιτυχία σας το λέω διπλά και τριπλά έτσι ώστε να διευκολύνετε και εμάς. Όσον αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα, είμαι εισηγητή για το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την Ελληνική Προεδρία ε, για την ε, συνεργασία και την καλή διάθεση συνεργασίας που έδειξε μέχρι τώρα. Ε, συμμερίζομαι λοιπόν τον, ε, τον προσεκτικό ε, ενθουσιασμό και την προσεκτική αισιοδοξία του ε, κύριου Υπουργού. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε να καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια έτσι ώστε να μπορέσουμε να πιέσουμε λίγο και το Συμβούλιο μέχρι το Μάρτι να έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Θα πρέπει να δουλέψουμε κυρίως με τρόπον ώστε να ε, οριμάσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα ε, και οι τεχνολογίες που άλλωστε έχουν αναπτυχθεί ήδη να οριμάσουν οι καταστάσεις ε, και στον ιδιωτικό τομέα. Ξέρετε ότι όσον αφορά το φυσικό αέριο και το υγροποιημένο και το άλλο έχει τεχνολογίες οι οποίες είναι ήδη ιδιαίτερα προχωρημένες. Επίσης και το θέμα των εκπομπών μας ενδιαφέρει πολύ στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Οπωσδήποτε όμως αυτή η πρόταση δεν θα πρέπει πρέπει να απογυμνωθεί ε, ε, λόγω των targets που, έχουμε, που έχουν μπει. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει οι στόχοι να είναι, να είναι ρεαλιστικοί, αλλά φυσικά θα πρέπει να υπάρχουν γιατί δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε ομοιογένεια του δικτύου σε ευρωπαϊκό επίπεδο και άλλωστε γι' αυτό αποφασίσαμε να κάνουμε κάτι για να υπάρχει η ομοιογένεια και κάτι άλλο όσον αφορά τα θέματα τουρισμού, έστω και αν δεν είναι απολύτω δικιά σα αρμοδιότητα, το ξέρω αυτό, ελπίζω ότι θα μεταφέρετε το θέμα στον ε, αρμόδιο καθήλη Υπουργό. Μα ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα τουριστικά ε, ζητήματα. Ελπίζουμε ότι τον ε, Μάρτιο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει την απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ελπίζουμε ότι στη διάρκεια τη ελληνική προεδρία θα ξεκινήσει αναθεώρηση των κωδίκων όσον αφορά τη τις ε, θεωρήσεις ε, και ελπίζουμε να ε, ετοιμάσετε τον δρόμο και για μας. Ξέχασα να σας χρονομετρήσω, αλλά δεν πειράζει. Ο κύριος Μαρινέσκου, δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ. Ακούσατε και τους συναδέλφους μου. Εγώ είμαι εισηγητής για τον ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Ακούσατε και τα σχόλια των σοσιαλιστών, αλλά και οι φιλελεύθεροι και το ΕΛΚ. Το ίδιο πράγμα σας ζητά να ε, θίξετε το θέμα του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Εδώ θα έχουμε στην Επιτροπή και ψηφοφορία, επομένως θα έχετε και την ε, θέση του Κοινοβουλίου. Το μόνο που σας ζητώ είναι να κινήσετε τις συζητήσεις. Ξεκινήστε τη συζήτηση. Μην ακούτε τους συμβούλους που σας λένε ότι είναι αδύνατον. Εγώ αλλά γενικά, εμείς εδώ θεωρούμε ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει συμφωνία, συμβιβασμός ε, με το Συμβούλιο. Θα έχετε το κείμενο της Επιτροπής και νομίζω ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Αυτό είναι το δικό μου αίτημα λοιπόν, η δική μου έκκληση. Ξεκινήστε τις συζητήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, πριν ε, σας ε, δώσω και πάλι το λόγο, ένα σημαντικό θέμα που ήθελα να θέξω εγώ ως Πρόεδρος είναι το ζήτημα των πακέτων για τους υδροδρόμους του πακέτου για του σιδηροδρόμου ε, και βλέπω ότι θέλετε πραγματικά να προχωρήσει αυτό το πακέτο, ιδιαίτερα στην τεχνική του πτυχή. Εμείς θα ψηφίσουμε για, επί του συνόλου του πακέτου το Φεβρουάριο. Είμαστε θετικά διακείμενοι, ανοιχτοί, να εξετάσουμε τα τεχνικά ζητήματα ξεχωριστά για να σημειωθεί πρόοδος πριν από το τέλος της ε, θητείας μας. Επικρατώ λοιπόν τα όσα είπατε, γιατί λαμβάναμε κάποια αρνητικά μηνύματα ότι το Συμβούλιο δηλαδή δεν θα το εξετάσει καθόλου. Και υπήρξε μια αναταραχή στα μέλη του Κοινοβουλίου που μπορώ να σας πω. Το άλλο που ήθελα να θίξω είναι ο κανονισμός 261 για τα δικαιώματα του πιβάτη του ε, κυρίου Μπαχ. Ο τίτλος είναι δικαιώματα του επιβάτη, των επιβατών και όχι των αεροπορικών αερογραμμών. Των επιβατών λοιπόν τα δικαιώματα και θα έπρεπε να υπενθυμίσετε και στα μέλη, κάποια μέλη του Συμβουλίου ότι πρόκειται για δικαιώματα του επιβάτη και όχι των αεροπορικών εταιριών. Κύριε Υπουργέ. Thank you, Mr. Simpson. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σίμψον. Βουλευτές, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ε, τόσο μεγάλη συμμετοχή στη συζήτηση και την... το γεγονός ότι θίξατε μια σειρά από πολύ σημαντικά θέματα <clears throat> που αφορούν ε, τον τομέα τον οποίο εκπροσωπώ ως ε, Προεδρία του τομέα των μεταφορών. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το κεντρικό ζήτημα το οποίο θέσατε όλοι. Το ζήτημα του σιδηροδρομικού πακέτου. Θέλω να σας πω και θέλω να σας διαβεβαιώσω και θέλω να εκφράσω με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο την πολιτική μου βούληση και την πολιτική μου απόφαση ως πρόεδρος του Συμβουλίου ότι θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ολοκλήρωση αυτού του πακέτου. Πριν από λίγο συνάντησα και τον <coughs> Αντιπρόεδρο και Επίτροπο, τον Αρμόδιο Επίτροπο, τον κύριο Κάλλας, με τον οποίο ε, μάλιστα είναι πάρα πολύ αποφασισμένος, φιλόδοξος και αποφασιστικός ό,τι αφορά την προώθηση του πακέτου. Αποφασίσαμε λοιπόν, επειδή αυτό το πακέτο είναι πάρα πολύ, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ και δυστυχώς δεν έχουμε εμείς ως ελληνική προεδρία καμιά ευθύνη για αυτή την καθυστέρηση, αποφασίσαμε λοιπόν από κοινού το Συμβούλιο, η Επιτροπή και παρακαλώ ε, κύριε Πρόεδρε και εσάς, την Επιτροπή σας, μέσα από τους ε, επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων ε, και τους ραπορτέρ, να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια, ώστε να καταβληθεί από όλους μια κοινή προσπάθεια να οργανωθεί ένα timeline, ένα οργανόγραμμα, ένα χρονοδιάγραμμα, έτσι ώστε να δούμε αν μπορούν να χωρέσουν όλες αυτές οι δραστηριότητες το επόμενο χρονικό διάστημα εάν χωράνε και είναι υλοποιήσιμο, υλοποιήσιμη αυτή η διαδικασία, εγώ θα είμαι εδώ κάθε μέρα ως πρόεδρος του Συμβουλίου για να κάνω και κάτι άλλο. Ε, δυστυχώς, επειδή με ρώτησε κάποιος συνάδελφος, η συντριπτική πλειοψηφία των, ε, μελών, των κρατών μελών του Συμβουλίου είναι από αδιάφορη έως αντίθετη στο πακέτο αυτό στην πρόοδο αυτού του πακέτο. Υπάρχει και αυτός ο παράγοντας δηλαδή που πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι δεν υπάρχει προθυμία από τα κράτη-μέλη να προχωρήσει αυτό το πακέτο σε αυτόν τον χρόνο τον ασφυκτικό λέγοντάς μας, τουλάχιστον εγώ αυτά τα μηνύματα πήρα από συναδέλφους μου τις τελευταίες μέρες που επικοινώνησα με κάποιους από αυτούς, μην προχωρώ, προχωράτε αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Τα δύο θέματα, όπως, πολύ καλά ξέρετε, έχουν κλείσει. Έχει απομείνει το ένα, το ζήτημα του ERA και αυτή την προσπάθεια θα κάνουμε. Υπόσχομαι λοιπόν εδώ ενώπιόν σας και δεσμεύομαι ότι το επόμενο χρονικό διάστημα σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή θα καταβάλουμε όλη μας την προσπάθεια προκειμένου να προχωρήσει και να ολοκληρώσουμε και αυτό το πακέτο. Αυτό είναι μια καθαρή δήλωση που θέλω να κάνω ενώπιον σας, έντιμη πολιτική δήλωση, την οποία εννοώ και θα καταβάλω κάθε προσπάθεια και θα ξανάρθω στην Επιτροπή να σας πω και πώς προχωρούν οι διαδικασίες. Αλλά απλά επαναλαμβάνω υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα της Προεδρίας μας που ουσιαστικά στα μέσα Μαρτίου διακόπτονται οι εργασίες του Κοινοβουλίου. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα του shift to rail θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία η οποία έρχεται να ενώσει σε μια πολύ βαθιά συνεργασία τη βιομηχανία, την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την ευρωπαϊκή σιδηροδρομική βιομηχανία τα πανεπιστήμια, τα Ινστιτούτα, τα ερευνητικά ιδρύματα, τα κράτη-μέλη σε μια κοινή προσπάθεια για να αναπτύξουμε τα επόμενα χρόνια σε ένα υψηλό τεχνολογικό βαθμό προς το καλό της ανάπτυξης της Ευρώπης και των επιβατών, των Ευρωπαίων πολιτών, το, το σιδηρόδρομο στην Ευρώπη. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να κλείσουμε το ζήτημα στις 14 Μαρτίου στο Συμβούλιο προκειμένου να προχωρήσουμε στη συνέχεια για να γίνει και ο κανονισμός του Συμβουλίου με σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα προσπαθήσω πολύ γρήγορα να απαντήσω και στα επόμενα ερωτήματά σας ε, πολύ τηλεγραφικά και θα προχωρήσω και σε άλλες λεπτομέρειες στη συνέχεια. Σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά κάψιμα, πάει πάρα, πάρα πολύ καλά ο φάκελος αυτός. Ο τελευταίος τρίλογος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα γίνει στις 5 Μαρτίου και κλείνουμε. Τα αεροπορικά, στα αεροπορικά, τα δικαιώματα των επιβατών, ε, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Σίμψον πριν από λίγο, να αναφερθούμε σε αυτά, να δώσουμε την προσοχή μας, το επίκεντρο της πολιτικής μας προσπάθειας στα δικαιώματα των επιβατών, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι ένας, ακριβώς για αυτό το λόγο, είναι ένας εξαιρετικά ευαίσθητος και δύσκολος φάκελος. Δεν έκλεισε στη Λιθουανική Προεδρία. Ο στόχος είναι να κλείσουμε, να τον κλείσουμε το αργότερο στις 5 Ιουνίου στο Συμβούλιο που θα γίνει. Σε ό,τι αφορά το e-call θα κλείσει μέχρι το Μάρτιο. Εξαρτάται βέβαια όπως ξέρετε και από έναν άλλο φάκελο που ανήκει σε ένα άλλο Υπουργείο στην, στην Προεδρία μας, σε ένα άλλο Συμβούλιο εννοώ, στο το Συμβούλιο του Υπουργείου ε, Ανάπτυξης που έχει σχέση με τις προδιαγραφές των συσκευών. Ελπίζω λοιπόν να κλείσει και αυτό, ούτως ώστε να πάμε όλοι μαζί. Σχετικά με το ζήτημα, σχετικά με το ζήτημα των σλότς που έθεσαν κάποιοι συνάδελφοι. Από το πακέτο του αεροδρομίου εμείς έχουμε δώσει προτεραιότητα στην πρόταση για το θόρυβο. Είμαστε πρόθυμοι για τις άλλες δύο προτάσεις αλλά όπως καταλαβαίνετε τα χρονικά περιθώρια είναι πάρα πολύ στενά για τη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε κάθε περίπτωση θα προχωρήσουμε στη συζήτηση στο επίπεδο του Συμβουλίου. Για τα δικαιώματα των επιβατών επανέρχομαι. Η Ελλάδα έβαλε αρχικά τη διαπραγμάτευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι τυχαία. Ακριβώς για το λόγο που είπε προηγουμένως ο κύριος Πρόεδρος, ο κύριος Σίμψον. Γιατί θέλουμε να δώσουμε έμφαση όπως και εσείς τονίσατε, στα δικαιώματα και στην στήριξη και στην προστασία των επιβατών. Εφόσον θα είχε επιτευχθεί συμφωνία στο Συμβούλιο της ε, Λιθουανικής Προεδρίας δεν έγινε με πολλά εκκρεμή ζητήματα με αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα αριθμό προβλημάτων που δεν έχουν επιληθεί εάν προσθέσουμε και το περιορισμένο διάστημα της τρέχουσας νομοθετικής περίοδου ε, πιστεύω ότι και φιλοδοξώ ότι θα μπορέσουμε στο, όπως είπα προηγουμένως, το τελευταίο συμβούλιο να το περάσουμε. Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός. Σημαντική πρόταση, έχει υποστηρικτές, αλλά έχει και επικριτές όπως ξέρετε έχει και εγωισμούς θα έλεγα όπως είπε ο κύριος Δανέλης προηγουμένως ειδικά στο Συμβούλιο ανάλογα με την εξέλιξη των θεμάτων που έχουμε ως προτεραιότητα και το διαθέσιμο χρόνο θα προχωρήσουμε στην εξέτασή του. Σε ό,τι αφορά το Connecting Europe Facility θα συνεργαστούμε με την Επιτροπή και όλους τους ε, Ευρωπαίους συντονιστές σχετικά με τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Θέλουμε να συνεργαστούμε την Επιτροπή και τους συντονιστές. Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου, αφού θεωρώ ότι συνδέεται στενά με την ανάπτυξη και την πρόοδο. Η συντονισμένη ανάπτυξη υποδομών για όλα τα μέσα, σιδηρόδρομος, δρόμοι, λιμάνια κλπ. είναι ζωτική σημασία για την Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να τονίσω ορισμένες σημαντικές παραμέτρους συμπληρώνοντας όσα είπε ο κύριος Κουμουτσάκος και συμφωνώντας μαζί του θα ήθελα όμως να συμπληρώσω και να σας θυμίσω ή να σας ενημερώσω για όσους ε, δεν γνωρίζουν ότι ως υπουργό ε, Υποδομών τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα είχα μια εμπειρία γιατί ξεκινήσαμε, επανεκκινήσαμε ως κυβέρνηση τους αυτοκινητόδρομους που ήταν ε, project μικτά με ιδιώτες, με τράπεζες και το, το δημόσιο, βασικά με ευρωπαϊκούς πόρους, με μια μεγάλη στήριξη, οφείλω να το πω, και να το τονίσω και να ευχαριστήσω με μια πολύ μεγάλη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των οργάνων της, μπορέσαμε και ξαναβάλαμε μπροστά ένα μεγάλο project αξίας περίπου 7,5 με 8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο υπάρχουν ορισμένες εμπειρίες από αυτήν την προσπάθεια που κάναμε που θέλω να σας τις περιγράψω και κυρίως έχει να κάνει με το τραπεζικό τομέα ο οποίος συμπεριφέρεται με πολύ μεγάλη σκληρότητα χωρίς καμία, καμία ευελιξία Επίσης θέλω να σας τονίσω και να σας αναφέρω ότι ακόμα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η οποία έχει το, το γνωστό AAA και δεν πρέπει να το χάσει συμφωνούμε αλλά από την άλλη πλευρά είναι ο οργανισμός ο οποίος, ο τραπεζικός οργανισμός, το πιστοτικό ίδρυμα που πρέπει να βοηθήσει την Ευρώπη να αναπτυχθεί γιατί αν δεν υπάρξουν δημόσιες επενδύσεις μαζί με τις ιδιωτικές είναι δύσκολο να αναθερμανθεί η οικονομία στην Ευρώπη και κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν υποστεί πολύ μεγάλο πλήγμα από την κρίση όπως είναι η Ελλάδα και όχι μόνο. Συνεπώς κάνω έκκληση να γίνει μια συζήτηση οργανωμένη σχετικά με το πώς όλο αυτό το δίκτυο το οργανωμένο που πρότεινε προηγουμένως ο κ. Κουμουτσάκος τα ευρωπαϊκά δίκτυα να ενταχθούν σε ένα συνολικό πρόγραμμα για το οποίο θα αρχίσει μια σοβαρή χρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αποφάσεις του Συμβουλίου αλλά κυρίως από τον τραπεζικό τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν και ιδιώτες. Αυτό νομίζω ότι αποτελεί, αυτό νομίζω ότι αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη συνολικότερα στην Ευρώπη. Ε, σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά κάψιμα επανέρχομαι και λέω ότι θα το τελειώσουμε στις 5 Μαρτίου. Σε ό,τι αφορά, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που έχουν να κάνουν επαναλαμβάνω με το θέμα των ε, βαρών και των ε, διαστάσεων θα ήθελα να πως τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν αγωνίες από ορισμένε χώρες ότι θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε μία ισορροπία ανάμεσα στα, στις ανησυχίες αλλά και στα ζητούμενα ούτως ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω επιβαρύνσεις στους δρόμους ορισμένων χωρών που είναι χώρες διέλευσης. Από την άλλη πλευρά όμως οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου να ενισχύσουμε την κίνηση αυτοκινήτων με απεξάρτηση από το πετρέλαιο, ηλεκτρικά δηλαδή αυτοκίνητα, ε, έτσι ώστε να γίνουμε πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, αλλά και να δημιουργήσουμε μέσα από την ανάπτυξη αυτών των αυτοκινήτων ε, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη της τεχνολογίας. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της εσωτερικής ναυσιπλοείας, θεωρώ ότι είναι κρίσιμο ζήτημα και θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε ούτως ώστε στον κανονισμό, ότι, ώστε ο κανονισμός να εγκριθεί από το Συμβούλιο του Ιουνίου. Αυτές είναι οι απαντήσεις μου σε όλα τα ερωτήματα τα οποία θέσατε. Θα προσπαθήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να γεφυρώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών μέσα στο Συμβούλιο, των ε, κρατών μελών και του Κοινοβουλίου, ώστε όλες οι προτάσεις να μπορούν να έχουν μια τελική μορφή, να είναι φιλόδοξες και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Ευρώπης και των πολιτών της, έτσι ώστε μέσα από τις ισορροπίες που αναγκαστικά έχουν αυτές τις αποφάσεις, κυρίως να οδηγηθούμε στο να ενισχύσουμε μια αρετή που πρέπει να διακρίνει την πολιτική. Και η αρετή που πρέπει να διακρίνει την πολιτική δεν είναι άλλη από το να είναι αποτελεσματική και χρήσιμη για τους πολίτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much indeed, Minister. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσίασή σας βεβαίως και για τις απαντήσεις που δώσατε στις ερωτήσεις των βουλευτών. βλέπουμε στη συνεργασία μαζί σας, όπως είπατε, όπως είπε και ο προκάτοχός σας, μπορεί το Κοινοβούλιο να κλείνει τον Απρίλιο ή όποτε κλείνει, η περιπτώσει. Πρόεδρος είμαι έως την 1η Ιουλίου. Θα είμαι λοιπόν πάντα στο πλευρό σας αυτή την Προεδρία. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε ασφαλώς στα θέματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως, όπως άλλωστε ακούσατε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω στην καλή συνεργασία για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Okay, guys, can we go on to... Παρακαλώ. Να συνεχίσουμε λοιπόν. Ένα τελευταίο έχουμε στην ημερήσια διάταξη σημείο. Μέγιστε επιτρεπόμενε διαστάσεις σε διεθνεί και εθνικές μεταφορές. Έχουμε 65 τροπολογίες. Δεν ξέρω αν ο εισηγητής ε, μπορεί να πει ότι ε, είναι τόσες πολλές αυτές που ασχολούνται, που αφορούν μάλλον το διαστηνοριακό ε, εμπόριο και μεταφορές μάλλον. Κύριε Λάιχτφριντ, κύριε Λάιχτφριντ λέω, μήπως θα μπορούσατε να πάτε προς τα έξω σιγά σιγά και τα πηγαδάκια να τα κάνετε έξω, έτσι ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Γιώργ Λάιχτφριντ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, την συνάδελφοι. Έχουμε την έκθεση αυτή σε μια φάση όπου έχει ολοκληρωθεί ένα μέρος του έργου, αλλά το άλλο έχει μείνει και περιμένει. Αυτό που έχει ολοκληρωθεί είναι οι αρχικές θέσεις που εκφράζουν οι συνάδελφοι. Ξέρουμε δηλαδή ο καθένας τι θέλει, που τοποθετείται, πώς εκφράζεται, αλλά ίσως θα μπορούσαμε να αξιολογήσουμε και τις πιθανές πλειοψηφίες ανάλογα με τις διάφορες ε, ψηφοφορίες που μπορεί να γίνουν, πώς μπορούν να διαμορφωθούν αυτές οι, οι και προσπαθώ έτσι να ε, κάνοντας αυτήν την αξιολόγηση να υπολογίσω και τους, τα σημεία μπορεί να έχουν πιο πολλές δυσκολίες για να τα περιορίσω. Τε, δύο τομείς λοιπόν βλέπω, κυρίως ε, στην ουσία αυτών των τροπολογιών. Τέσσερις τομείς λοιπόν διαφορετικούς, τρεις σχετικά ε, μη προβληματικούς και υπάρχει και το θέμα των αεροδυναμικών μέτρων όπου οι τροπολογίες των συναδέλφων ε, ανάλογα με μήκος και όλα τα υπόλοιπα τεχνικά στοιχεία διαφοροποιούνται αρκετά. Έχουμε μια πρώτη συζήτηση, πραγματοποίηση με τους και ηγητές που δείχνει νομίζω ότι έχουμε προχωρήσει αρκετά για να βρούμε λύσεις στον τομέα αυτών που μπορούν να ε, υποστηρίξουν στον δυνατόν περισσότεροι συνάδελφοι με μεγάλη πλειοψηφία. Το ερώτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί ή πόσο μπορεί να ε, αυξηθεί το μήκος του φορτηγού ε, προς τα μπρος για να γίνει πιο ενοδυναμικό. Μιλάμε για 400 με 800 μιλιμέτρα. Τα flaps επίσης και το θέμα της σύγκρουσης ή αποφυγής καλύτερα σύγκρουσης αυτών των μέτρων με υφιστάμενες διατάξεις ευρωπαϊκές ή διεθνείς. Και βέβαια, ε, ό,τι μέτρα θα εισαγάγουμε θα, θα πρέπει να φέρουν σε δυσμενέστερη ανταγωνιστική θέση τη δική μας βιομηχανία. Ένα άλλο ζήτημα λοιπόν είναι αυτό τη αύξηση του βάρους λόγω των εναλλακτικών ε, συστημάτων όθησης. Έχουμε συζητήσει αρκετά, έχουμε προχωρήσει επίσης. Ο τρίτο τομέα είναι αυτός της ασφάλειας που δεν μπορούσαμε να συζητήσουμε σήμερα, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε ε, να περιμένουμε ευρύτερη υποστήριξη στην ε, βελτίωση της ασφάλειας των φορτηγών τόσο έξω από τις πόλεις όσο και μέσα στις πόλεις όπου έχουμε τα πιο πολλά ατυχήματα με θύματα ε, όπου εμπλέκονται φορτηγά. μία λύση ενδεχομένως να είναι να υπάρχει ένας ε, μετρητής βάρους, ένας δείκτης βάρους. Αυτή είναι η δουλειά στην οποία θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Και θα αναφέρω και ένα πέμπτο τομέα, ο οποίος μπορεί να έχει μεγαλύτερη βαρύτητα συναισθηματική, συγκινησιακή και ενδιαφέρον για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπου παρουσιάζεται και μια σειρά από αποκλίνουσες απόψεις. Έκανε ε, μια πρόταση η Επιτροπή, η οποία είναι πολύ ριζοσπαστική, πολύ ριζική, δεν βαίνει προς την αρθή κατεύθυνση και η δική μου η απάντηση ήταν εξίσου ριζική. Αντιδιαμετρικά αντίθετες λοιπόν, διαμετρικά αντίθετες λοιπόν οι δύο θέσεις. Και αντίστοιχα βλέπουμε και τις προτάσεις με τις τροπολογίες των συναδέλφων ανάλογα με τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πιστεύουν ότι το άνοιγμα των ορίων για τα μεγαλύτερα και βαρέα φορτηγά είναι και καλό και χρήσιμο. Ε, υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε, αλλά ρωτάνε το πώς και δεν θα πρέπει να υποχρεωθεί κανείς να δεχθεί ε, βαρέα ή πολύ μεγάλα ε, φορτηγά στη, στη χώρα του, άρα θα πρέπει να ισχύουν εθνικοί κανόνες. Και υπάρχει πέραν αυτού και Μία πρόταση που λέει αν πρέπει να γίνουν ανάμεικτες ε, λύσεις με ιδιαίτερες ρυθμίσεις ενώ κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν πρέπει ποτέ να επιτραπούν τα πολύ βαρέα, τα πολύ μεγάλα φορτηγά. Πρέπει λοιπόν να βρούμε λύσεις εδώ μέσα αυτές τις ε, αντίθετες απόψεις. Θέλω να πω το εξής, ότι εφόσον η λύση είναι να προχωρήσουμε με βάση τις ε, προτάσεις που ασκούνται και τις πιέσεις που ασκούνται, θα πρέπει να ακολουθήσουμε μέτρα τα οποία δεν έχουν προσβληθεί. Εκεί όπου ισχύει το μέτρο, στην Βόρεια Ευρώπη, την Ιρλανδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί όπου παίζει κάποιο ρόλο το μήκος ή το ύψος ή το βάρος, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία ή την Βόρεια Ευρώπη, τότε θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το περιθώριο να συνεχίσουν τα κράτη ε, όπως το επιθυμούν. Εφόσον βρούμε συμβαστική λύση. Εάν όμως δεν βρούμε συμβαστική λύση, τότε τα πράγματα θα είναι δύσκολα γιατί οποιοδήποτε μέτρο ισχύσει θα ισχύει για όλους. Γι' αυτό ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε συμβαστική λύση. Κάναμε καλές συστήσεις σήμερα. Δεν είναι σαφές το προς τα ποια κατεύθυνση θα προχωρήσουμε. ελπίζω όμως η Επιτροπή να μας προσφέρει την υποστήριξή της για τις προσεχείς εργασίες μας. Η κατάσταση είναι όπως την περιγράφω και περιμένω να ακούσω και τους συναδέλφους και βέβαια να παρακολουθήσω μια ενδιαφέρουσα και εντατική ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάιτφρίντε. Έχω χιλιομετρικό κατάλογο ομιλητών. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να είστε όσο γίνεται πιο λακωνικοί. και ε, δεν χρειάζονται όλοι να πούνε τα πάντα. Εάν το έχει πει κάποιος άλλος συνάδελφος, μην ε, αποφασίσετε να το πείτε κι εσείς. Ε, θα ξεκινήσουμε με τους Σκιώδης και μετά Κοκ, Μάισνερ, Φιώνα και έχουμε και την κυρία Τικάου και τον κύριο Φρίκο. Θα κλείσω τώρα τον κατάλογο των αγορητών. Όποιος πρόλαβε, πρόλαβε. Okay. Going, going. Και μην ε, σηκώνει ο καθένας το χέρι του τελευταία στιγμή, ε, θέλω και εγώ να μιλήσω. Τελείως έκλεισε ο κατάλογος. Κύριε Πρόεδρε, λέει ο κύριος ε, Σαρβάμα, όσον αφορά τώρα μια γενική σκέψη ή έναν έτσι συνολικό στόχο αυτής της νομοθεσίας, αν υπάρχει κάτι τέτοιο, θα είναι ότι θα πρέπει να είναι η νομοθεσία αυτή σαφής και συνεκτική. Αυτό περιμένουν όλοι από εμά και η αυτοκίνητο βιομηχανία και ε, αυτοί που ασχολούνται με τις εταιρείε μεταφορών και οι οδηγοί και οπωσδήποτε και οι πολίτες των κρατών μελών, των οποίων δηλαδή η οικονομία ε, και των οποίων οι θέσεις απασχόλησης ε, εξαρτώνται από αυτές τις αποφάσεις. Χρειαζόμαστε λοιπόν σαφήνεια και ε, συνέπεια, συνέχεια. Επί της ουσίας υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και αναφέρομαι σε αυτούς. Είναι περιβαλλοντικά ε, και οικονομικά βιώσιμα οχήματα. Φορτηγά που να καλύπτουν λοιπόν και την περιβαλλοντική και την οικονομική διάσταση και νομίζω ότι μπορούμε να το επιτύχουμε. Δεν βλέπω πολλά προβλήματα. Στις τροπολογίες τώρα, αν θα έχουμε 600 ε, μιλιμέτρα ή λιγότερο, αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Μη χάνουμε, μη σπαταλάμε χρόνο για αυτές τις λεπτομέρειες. Κάτι άλλο. Πιο ασφαλή φορτηγά. Και αυτό μπορεί να γίνει. Υπάρχει ήδη αρκετή τι συνένεση γι' αυτό. Νομίζω ότι έχουμε δει και κάποιες, κάποιους συμβιβασμούς επ' αυτών. Τώρα το θέμα αυτό το διασυνοριακό. Ε, δεν θα αναφερθώ μακρόν στο θέμα αυτό τούτη τη φορά, αλλά αναρωτιέμαι. Και μάλιστα εδώ παρεπιπτόντας να πω ότι ευχαριστώ και τον εισηγητή τον κύριο Λάιχτφριντ για την ε, πολύ εξαντλητική δουλειά που έκανε για το θέμα αυτό. Ωστόσο, αναρωτιέμαι, εκεί που είπατε ότι υπάρχουν τέσσερες κατηγορίες όσον αφορά ε, το διασυναριακό κομμάτι, ε, αυτές οι τρεις από τις τέσσερις όμως μου φαίνονται ταυτόσιμες με πολύ μικρή διαφορά δηλαδή αν μιλάμε για τη Φιλανδία προς τη Σουηδία ή αν έχουμε ε, τροπολογίες οι οποίες ε, ξεκινάνε από χώρες οι οποίες έχουν δοκιμαστικές περιόδους, Βέλγιο, Δανία, κάτω χώρες που νομίζω ότι ε, ήδη έχουν ολοκληρώσει τα των δοκιμαστικών περιόδων από το 2011. Ε, και μετά έχουμε και αυτό το, αυτό το διάδρομο Μπένιον, αλλά αυτό είναι το τρίτο σκέλος. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι όλα αυτά μας οδηγούν ε, στο να δεχτούμε το γεγονός ότι εν τέλει τα σύνορα δεν μπορούν να κλείσουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό και θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Thank you, Mr. Benyon Corridor. Κύριε Μπένιον που έχετε και δικό σας διάδρομο στο όνομά σας. Ναι, ναι, το δέχομαι, το δέχομαι. Είναι δικιά μου ιδέα. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω, Πρόεδρε, που μου δώσατε το λόγο και να ευχαριστήσω και τον Γιώργο γιατί δούλεψε πολύ σκληρά για το θέμα αυτό και συνεργάστηκε πολύ καλά μαζί μας ε, στην έκθεση αυτή. Όπως είπε μόλις και ο κύριος Σάρμα, Είμαι πεπισμένο ότι θα βρούμε συμβιβασμού στα περισσότερα σημεία τα οποία συζητήσαμε πολλές φορές και τα ξανασυζητούμε και σήμερα. Υπάρχουν και κάποια σημεία βέβαια επί των οποίων θα πρέπει να θέσουμε τις σωστές παραμέτρους επί των οποίων θα πρέπει να επικεντρωθούμε. Π.χ. να παραμείνουμε εστιασμένοι σε κάποιες επιπλέον διαστάσεις οι οποίες θα κάνουν τα φορτηγά ασφαλέστερα και πρασινότερα. Χωρίς βέβαια να καταλήξουμε σε μια shopping list με μια σειρά στοιχείων που θα λένε πώς μπορούν ακριβώς τα φορτηγά να γίνουν πιο βαριά, πιο μακριά. Ας πούμε, εάν ε, ε, βάλουμε ε, επιπλέον χώρο για, τις, για τα ρημουλκά, για, για τα στοιχεία των ρημουλκών, αυτά βεβαίως δεν θα μπορέσουν να έχουν καμία ενεργειακή αποτελεσματικότητα. Τώρα, εάν ε, θέλουμε πραγματικά να λύσουμε ζητήματα συνολικά και ομοιογενώς, θα πρέπει να λύσουμε και τα ζητήματα της ομοιογένειας των δρόμων ε, και να λέμε ποιοι θα είναι οι διάδρομοι που θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς στις μεταφορές. Εναλλακτικά καύσιμα. Ανταυτού θα ήθελα να δω τεχνολογίες χαμηλής εκπομπής ε, ρήπων και διοξιδίου του άνθρακα Επίσης θα ήθελα να δω τα στοιχεία αυτά τα οποία ε, αφορούν την ε, χρήση βελτιωμένης τεχνολογίας ε, όσον αφορά την υπέρβαση την υπέρβαση συνολικού μήκους δια της προσθήκης αεροτομών. Δεν βάλανε από την Επιτροπή ε, όρια, το αποφάσισαν να αφήσουν εμάς ε, να το δούμε το θέμα αυτό. Ε, νομίζω ότι υπάρχει έτσι σχετική έρευνα και πιστεύω ότι χωρίς μεγάλες δυσκολίες θα φτάσουμε σε συμβιβασμούς και εδώ. Δεν μπορώ να στηρίξω τις τροπολογίες οι οποίες επιβάλλουν ε, κάποια συστήματα ε, ζυγοστάθμισης ε, με εργαλεία εντός του οχήματος. Κοιτάξτε, στην αντίθετη περίπτωση που προτιμώ εγώ, νομίζω ότι το δημόσιο χρήμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι λιγότερο και επίσης αντιμετωπίζουμε και το πρόβλημα της υπερφόρτωσης. Ε, βέβαια, εάν ε, τα μηχανήματα βρίσκονται στο όχημα, ε, τότε γίνεται πιο εύκολη η δουλειά για τους οδηγούς και για τη βιομηχανία, αλλά δεν μπορεί να είναι υποχρεωτική αυτή η αναφορά. Επίσης, πώς φτάνουμε σε αυτό το όριο του 1 προς, 200 χιλιό, προς 2.000 συγγνώμη, χιλιόμετρα για την φόρτωση. Ε, πώς φτάνουμε σε αυτό. Παρατήρηση εκτός μικροφώνου, οι διερμηνείς δεν ακούν. Θα τα δούμε αυτά με τους συναδέλφους. Ακόμα και με την Εύα, ακόμα και με την Εύα, ή, ακόμα και η Εύα λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι γι' αυτό. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, για πέστε τα τώρα εσείς. Ευχαριστώ. Όπως ξέρετε δεν είμαι υπέρ της κατάργησης όλων των ελέγχων. Είναι το μειονέκτημα που έχουν ορισμένα κρατημέλη. ότι δεν έχουν κανένας τύπου ελέγχους. Στους πολύ μεγάλους, με πολύ μεγάλες ε, αποστάσεις και μπορεί να κυκλοφορεί ένα όχημα για 800 χιλιόμετρα και να μην ε, ελεγχθεί ή να μην ελεγχθεί μέσα σε ένα χρόνο ολόκληρο. Ας είμαστε λοιπόν λίγο πιο σοβαροί με τους ελέγχους δεν έχουν μεταφέρει και δεν εφαρμόζουν σε εθνικό δίκαιο του ελέγχους, το, εθνικό, το ευρωπαϊκό δίκαιο, δηλαδή τα κράτη-μέλη και έτσι δεν είναι ούτε καν εξασφαλισμένε οι ελάχιστε προδιαγραφέ ασφαλείας. Α, ναι, όχι, με συγχωρείτε επειδή ήθελα να απαντήσω κατηδίαν, τώρα όμως θα μιλήσω γερμανικά. Στις επιμέρους τροπολογίες. Έχω κάποιες ε, επιφυλάξεις για τα εναλλακτικά καύσιμα στην καταγραφή των διαφορών κατηγοριών, ηλεκτρισμός ε, και άλλα. Ε, εξαρτάται από την διαδικασία παραγωγής. Όταν προέρχεται από την καύση του άνθρακα δεν έχουμε θετικό απολογισμό για τις κλιματικές αλλαγές και βέβαια για την πυρηνική ενέργεια ισχύει το ίδιο, αλλά για τις κλιματικές αλλαγές κατά κύριο λόγο ισχύει αυτό. Γι' αυτό λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να διατοδιπώσουμε κατά τρόπον ώστε να είναι σαφής η κατάσταση για τον πάροχο της ενέργειας. Δεύτερο σημείο που με ενδιαφέρει. Αυτή η ε, επέκταση του μήκου που μπορεί να εξασφαλίσει καλύτερε συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζομένους οδηγού κτλ. Δηλαδή την εισαγωγή αυτής τη κουκέτα και τα flaps βέβαια. Εάν συνολικά σημαίνει ε, αύξηση κατά ένα μήκο των μεταφορών, τότε βγαίνουμε από τι συνδυασμένε μεταφορές. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο δηλαδή. Άρα αυτό είναι πρόβλημα. Εκεί βλέπω τα τεχνικά προβλήματα. αλλά φαντάζομαι στην συνεδρία των συντονιστών και οδών εισηγητών μπορούμε να τα συζητήσουμε λεπτομερέστερα για όλα όσα έχουν να κάνουν με την διασυνοριακή διάσταση των μεταφορών. Πιστεύω ότι εάν ορίσουμε μια ούτως υπήν γεωγραφική έννοια που θα λέει να στο βορρά γίνεται αυτό αλλά όχι στο νότο ή κάποια κράτη μόνα τους δεν μπορούν να λάβουν την πρωτοβουλία κτλ. Νομίζω ότι νομικά θα έχουμε πρόβλημα, θα έχουμε λάτωμα. Γιατί θα οδηγεί σε διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με το κράτος μέλος. Πράγμα το οποίο γεννά πολλές δυσκολίες. Είναι άλλο το να μπορεί ένα κράτος αυτόνομα να λάβει κάποιες αποφάσεις. Είναι άλλη υπόθεση αυτή, άλλη περίπτωση. Αλλά το να λέμε ότι θα έχουμε μια πολλαπλή πρόταση η οποία θα ισχύει στο βορρά, δεν θα ισχύει στο νότο, θα ισχύει στις Άλπεις αλλά σε ορισμένες περιοχές ή δεν θα ισχύει καθόλου, τότε έχουμε διαφορετικές συνθήκες και γι' αυτό θα πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να επαληθεύσουμε τις νομικές ε, ε, προϋποθέσεις. Επίσης, μου φαίνεται πολύ επικίνδυνο το να ανοίξει μια τέτοια πόρτα το έχω πει πολλές φορές, ισχύει πάντα, διότι είναι δύσκολη περίσταση και αν τα κράτη εκείνα τα οποία έχουν αποφασίσει ε, για διαφορετικούς λόγους το καθένα να μην επιτρέψει την κυκλοφορία των mega trucks, των πολύ μεγάλων φορτηγών ε, ανεξάρτητος των λόγων για τον οποίο έχω αποφασίσει να μην τα επιτρέψουν, να υποστούν πιέσεις προκειμένου να ανοίξουν διαδρόμους, αυτοκινητοδρόμους και το καθεξής υποχρεωτικά μόνο και μόνο για να μπορέσουν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις να εξασφαλίσουν κάποια μικρά πλεονεκτήματα, εμένα αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ προβληματικό. Και επίσης ακούσαμε τις συνέπειες από την στρέβλωση του ανταγωνισμού για τις μικρότερες επιχειρήσεις, για την μετακύληση του κόστους σε επίπεδο κράτους. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι πρέπει τα κράτη να αποφεύγουν τα χρέη, δεν υπάρχει πια τόσο πολύ χρήμα. Πρέπει να το αποφεύγουμε λοιπόν αυτό να μετακυλίεται το ε, κόστος στο κρατικό προπολογισμό. Και θα ήμουν εν γέννη πάρα πολύ προσεκτική σε αυτή την υπόθεση, γιατί ανοίγουμε πόρτες που δεν θέλουμε και που μπορεί να μας φέρουν τα αντίξω αποτελέσματα, δηλαδή μέτρα κυρώσεων οικονομικών εις βάρος των κρατών εκείνων που δεν θα προτιμήσουν να ανοίξουν τους δρόμους και αυτοκινητοδρόμους τους ή που δεν θα τους, ε, διευρύνουν τους αυτοκινητοδρόμους τους έτσι ώστε να μπορούν τα πολύ μεγάλα φορτηγά, τα Megatrax να τους χρησιμοποιούν. Θα το δούμε αυτό μπροστά μας έτσι και συμβεί, έτσι και προχωρήσουμε σιγά σιγά θα το δούμε να συμβαίνει και νομίζω τελικά θα φτάσουμε σε συνθήκες απόλυτης ανισότητας μεταξύ των κρατών εκείνων τα οποία για λόγους γεωγραφικούς ή άλλους ή και γιατί ε, έχουν, αυτή, έχουν προβεί σε αυτήν την επιλογή, επιβάλλουν πιο αυστηρές διατάξεις και προδιαγραφές. Ε, θέλω να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτό το θέμα. Ξέρετε όλοι βέβαια ότι είμαι πάντα πολύ επιφυλακτική, γιατί όταν ε, ταυτόχρονα θέλουμε να προωθήσουμε τον ε, σιδηρόδρομο, αλλά και επιτρέπουμε την ανάπτυξη αυτού του πολύ πιο φθηνού ανταγωνιστικού μέσου των, μεγάλων, των πολύ μεγάλων φορτηγών, μάλλον δεν κάνουμε σωστή δουλειά. Αυτές λοιπόν τις επιφυλάξεις έχω εκφράσει πολλές φορές. Ο κύριος Βαντάλλας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Πρόεδρε, πρόκειται για μια εξαιρετική στιγμή. Οι οδικές μεταφορές ε, έχουν βρει μια εξαιρετική καινοτόμα ιδέα για το, με το Eco καλή για το περιβάλλον, καλή για τις ε, οδικές μεταφορές και εμείς το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να δώσουμε και τη δική μας ε, θέση για να προωθήσουμε και αυτό το τομέα πολιτικής. Μα πόσο πετυχημένοι είμαστε επιτέλους ε, και με όλα αυτά τα εξαιρετικά πολύ επιτυχημένα πειράματα τίποτα δεν μένει να γίνει, μπορούμε να τελειώνουμε πάρα πολύ γρήγορα. Ε, δεν θεωρώ καθόλου ριζοσπαστική την ε, πρόταση της Επιτροπής, είναι αρκετά αξισορπημένη, μπορώ να το πω αυτό, όμως νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε, είναι πολύ απλά τα πράγματα ο εισηγητής είπε ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που πρέπει να επιληθούν. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Μόνο ένα πρόβλημα, η παρέμβαση της κυρίας Λίχτεμπεργκερ, γιατί ακούγοντάς την και βλέποντας και τις τροπολογίες της, ε, τελικά θα έχουμε ένα king size κρεβάτι μέσα στο φορτηγό, αλλά για τα υπόλοιπα που μας ενδιαφέρουν πραγματικά δεν κάνουμε τίποτα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο. Διατηρούμε μόνο την έκκληση για τις δικές μας αντροπολογίε, τι οποίες εμεί θεωρούμε σωστές και τις οποίες στερίζουμε για την γενοτομία, να είμαστε ω δυνατόν πιο κοντά στην πρόταση τη Επιτροπής, να αφήσουμε κατά μέρο όλες αυτές τις περιττές λεπτομέρειες που φτάνουμε σε ε, απίστευτη λεπτομέρεια πολύ συχνά σε αυτό το κοινοβούλιο, σας παρακαλώ Πρόεδρε, δεν χρειαζόμαστε τέτοια εδώ. Ας μείνουμε κοντά στην πρόταση της Επιτροπής. Τώρα για το διασυναρικό εμπόριο να δώσουμε κάποιες ε, ευκαιρίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μενάλης. Βεβαίως θα ήταν θαύμα να συμφωνήσουν ECR ε, και πράσινοι σε αυτή την Επιτροπή. Κύριε Κόχ. Ναι, ευχαριστώ πρόεδρε. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι απογοήτευση. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο θέμα που να τη χάνει τέτοια ε, λαϊκιστική ε, και δημοσκοπική, δημοσκοπικής ε, κατάχρησης. Είναι τα φορτηγά που έχουμε αυτή τη στιγμή στους δρόμους μας ήδη πολύ επικίνδυνα για τις υποδομές, ε, για, τις, ε, για την κυκλοφορία είναι υπερφορτωμένα και δεν μπορούν να ε, σταματήσουν εγκαίρως όταν υπάρχει πρόβλημα. Άρα χρειάζεται οπωσδήποτε να προχωρήσουμε με πιο καλές διατάξεις. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τα μεγαλύτερα σε μήκος φορτηγά και για την ασφάλεια και για την αποτελεσματικότητα και για τις οδικές μεταφορές. Είναι μικρά βήματα οι αλλαγές στο χώρο της καμπίνας. Χρειάζονται πολύ περισσότερα πράγματα, ουσιαστική αναδιατύπωση του τι σημαίνει μεγάλο φορτηγό. Ευχαριστώ. Thank you, Mrs. Η κυρία Μάισνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή καθώς με τόση ψυχραιμία μας παρουσιάσει το θέμα αυτό, στο οποίο γνωρίζουμε ότι έχουμε σοβαρές αντιθέσεις απόψεων, όπου τα μέτρα, σταθμά, μήκη και πλάτη ε, να γεννήσουν μεγάλα πάθη. Πάντως μέλημα όλων μας είναι νομίζω να είναι ασφαλή τα φορτηγά, στα τέσσερα πρώτα σημεία δεν υπάρχει πρόβλημα, στο πέμπτο θα δούμε ότι θα υπάρχουν δυσκολίε για να συμβαστούμε, αλλά πάντως νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι εφόσον μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότητα και καινοτομία σε ένα είδο μεταφορών. Ε, διαλειτουργικά ναι, αλλά πάνω απ' όλα στόχο μα πρέπει να είναι η βελτίωση τη αποτελεσματικότητα και αυτό με την προκείμενη πρόταση, άλλωστε μα το έχουν δείξει και οι εμπειρίε μα από τα πιο μακριά και ογκώδη βεβαίως ε, φορτηγά μπορούμε να το εξασφαλίσουμε εφόσον υπάρχουν οι υποδομές τώρα για, την, ε, για τα όρια και την υπέρβαση ορίων. Ε, νομίζω ότι όπως ε, άλλωστε πάντα λέμε για την εσωτερική αγορά, έχουμε κοινό σύστημα μεταφορών. Το αναφέραμε και στις διευρωπαϊκές, στα ευρωδιευρωπαϊκά δίκτυα δεν μπορούμε να κάνουμε τα πάντα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε κάποια πράγματα διαφοροποιούμαστε και έτσι μπορεί σε κάποια πράγματα ένα κράτος μέλος να αποφασίζει αν διαθέτει τις υποδομές ή αν δεν τις διαθέτει και αν μπορεί ή δεν μπορεί να δώσει άδεια για κυκλοφορία στα, ε, στην επικρατεία του κάποιων πολύ μεγάλων φορτηγών. Εμείς και στη Βόρεια Γερμανία όπως ε, και αλλού Έχουμε σύστημα σοβαρό μεταφοράς των φορτίων με τις πλωτές οδούς. Δεν ζητούμε όμως από κανένα άλλο κράτος να αναπτύξει πλωτές οδούς το τις έχει. Γι' αυτό λοιπόν, εάν κάποια κράτη έχουν υποδομές τα οποία επιτρέπουν την αξιοποίηση μιας καινοτομίας τεχνολογία, τεχνολογικής, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να μπορούμε να το επιτρέψουμε αυτό. Και επίσης έχουμε κάνει μια τροπολογία μας με συναδέλφους η οποία στηρίζεται στην εμπειρία και τη γνώση από την ε, επιμελητία. Εάν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα για διμερείς επαφές, συζητήσει μεταξύ κρατών και περιφερειών που μπορούν να συμφωνήσουν ότι στην, ε, στις υποδομές, στο τάδε σημείο, από το τάδε έως το τάδε σημείο, στο τάδε διαδρομή, στον τάδε τομέα, μπορεί να ταξιδεύουν ε, περισσότερο τα πολύ μεγάλα φορτηγά, τότε γιατί όχι. Ε, έχουμε παραδείγματι και συστήματα τα οποία μπορούν να βελτιωθούν όπως αυτό το σύστημα συστήματος ε, πέδησης αλλά και κατάρτιση που μπορούμε να προσφέρουμε στους ε, οδηγούς, ειδική κατάρτιση. Αυτά στη Γερμανία προβλέπονται που μπορούν να επιτρέψουν την ασφαλή κυκλοφορία αυτών των πολύ μεγάλων φορτηγών. Δεν χρειάζεται να είμαστε όλοι ενάντια στην πρόοδο εάν θέλουμε να έχουμε ευρωπαϊκές μεταφορές. Κύριε Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να πω ότι πρώτη φορά έρχομαι στην Επιτροπή Μεταφορών. Δέκα χρόνια χρειάστηκαν, αλλά χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ μαζί σα, γιατί βεβαίω είχα κάποιε τροπολογίε και θέλω να, να παρακολουθήσω. Ε, σας έλεξαν τη βίζα όταν μπήκατε. Όχι, αυτά τα σύνορα είναι ακόμα ανοιχτά για να μπούμε στην αίθουσα. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Αλλά ήθελα να ακούσω και τα επιχειρήματα Είχα ανησυχήσει όταν διάβασα την έκθεσή σας. Συνήθως βεβαίως δεν ανησυχώ, αλλά τώρα που εσείς είπατε ότι πήρατε εξαιρετικά ε, ριζοσπαστική θέση, τώρα έτσι κάπως εξηγούνται τα πράγματα. Ε, βεβαίως που θα μπορούσε κάποιος να πει, εντάξει ξέρουμε ποια είναι η θέση του, είναι Σουηδός. Αλλά ουσιαστικά ασχολήθηκα με αυτό το θέμα γιατί είμαι και μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Έχω συνηθίσει τους συναδέλφους μου εκεί να παίρνουν μη ρεαλιστικές θέσεις σε ό,τι φορά τις μεταφορές. Να σας το πω πολύ ειλικρινά. Όμως με εξέπληξε το γεγονός ότι όταν έχουμε μια φιλική προς το περιβάλλον ε, λύση υπάρχουν επικρίσεις σε αυτή την Επιτροπή που δεν θέλει να εξετάσει αυτό το ζήτημα. Η πράσινη είναι κατά όλων των προτάσεων, ανεξαρτήτως ε, περιεχομένου. Αλλά εδώ σχόλιο εκτός μικροφώνου. Διακόπτει ο Πρόεδρο. Ε, όλα περνάνε από τον Πρόεδρο, συνάδελφοι. Συνεχίζει ο κ. Φέλνερ. Μόνο μία παρατήρηση. Θα ήθελα να καλέσω του συναδέλφου να μείνουν σε μία αρχή τουλάχιστον. Αποδέχομαι βεβαίω ότι κανεί δεν θα έπρεπε να του επιβληθεί να δεχθεί βαριά φορτηγά και μεγαλύτερα, μεγαλύτερου μήκου φορτηγά. Το κατανοώ. Αλλά να μην περιορίζετε και του υπόλοιπου που θεωρούν ότι μπορεί να υπάρξει λύση. Αλλά και μέσα στο εσωτερικό μια χώρα, αλλά και σε διαμετακόμιση και μεταξύ χωρών. Λοιπόν, δεν το επιβάλλουμε σε κανέναν, ούτε όμω να απαγορεύσουμε σε κάποιον να έχει αυτή την πεποίθηση. Αυτό θα μπορούσε να είναι πολύ καλή λύση για την οικονομία, για το περιβάλλον και για τον κλάδο αυτό τη βιομηχανία. Αυτή είναι η δική μου αρχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πολύ. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, όπως... Εδώ στα γερμανικά λέει ότι δεν θα πρέπει αυτό που ισχύει τώρα να υφίσταται πιέσεις. Αυτό είπε η κυρία Λιχτινπέργκερ, ότι θα πρέπει να πιέζονται αυτοί που έχουν ήδη ε, αυτή την ε, πρακτική στην Ιρλανδία, τον Ηνωμένο Βασίλειο, τι βορειέ χώρε. Ναι, και εγώ θα σα απαντούσα ότι δεν θα πρέπει αυτό να σχίσει ούτε για τη Γαλλία, ούτε την Αυστρία, ούτε για καμιά άλλη χώρα. Ωστόσο, έχουμε βέλτιστε πρακτικέ και με μεγάλη προσοχή τι συνεχίζουμε και στο μέλλον. Διότι δεν έχουμε παντού σιδηρόδρομο, δεν διαθέτουμε παντού πρώτε οδού. Εμείς από τι κάτω χώρε έχουμε εμπειρία με πολύ καλά και επιστημονικά στηριγμένα αποτελέσματα. Για τα όσα είπε η κυρία Μάιστερ, Μάιστερ και ο κύριος Κόχο, πιστεύω πρέπει πάνω απ' όλα να γίνει σεβαστή η αρχή της επικουρικότητας. Αυτό που προσπαθούμε πάντως με τις τροπολογίες μας είναι να καλύψουμε τις ανησυχίες κάποιων συναδέλφων που φοβούνται ότι θα γίνει δυνατή κυκλοφορία πολύ μεγάλων φορτηγών σε δρόμους όπου μπορεί να υπάρχει κίνδυνο φερρυπίν για τους ποδηλάτες. Εμείς από τι κατοχώρες έχουμε μεγάλη εμπειρία από ποδηλάτες και τους φροντίζουμε ιδιαίτερα και ξέρουμε πού θα πρέπει να πάνε αυτά τα μεγάλα φορτηγά. Κύριε Μπένιον, κύριε Μπένιον, εγώ σας συμπαθώ. Αλλά οι διάδρομοι Μπένιον καθόλου δεν μου αρέσουν. διότι δεν γίνεται σεβαστή επικουρικότητα στην περίπτωση αυτή. Γι' αυτό λοιπόν σας καλώ να αλλάξετε θέση στην υπόθεση αυτή και μαζί με τον κύριο Λάιχτφριντ με βέβαια ότι μπορούμε να βρούμε καλές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Foster. Κυρία Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα αποφύγω σχόλια τα οποία έγιναν ήδη και από τον οποίο πρέπει να βρεθεί λύση. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι εμείς μπορούμε να στηρίξουμε τις αλλαγές οι οποίες συζητιούνται, αλλά χρειαζόμαστε σαφήνεια όσον αφορά το σχεδιασμό. Ε, κάποιος μίλησε για ε, κρεβατοκάμαρα με διπλό κρεβάτι, τρεις ορόφους ή οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει αυτό. Όποιος και αν είναι ο σχεδιασμός, ε, και αυτό αφορά βέβαια και τους, την αυτοκίνητο βιομηχανία, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι μόνο το ύψος, το βάρος, το πλάτος, το μήκος, αλλά η ορατότητα, η μέγιστη δυνατή ορατότητα που πρέπει να έχει ο ε, οδηγός. Αυτό είναι ένα σημαντικό ζήτημα από το οποίο διαρκώς και αόκνος εργάζεται η αυτοκίνητο βιομηχανία. Ο σχεδιασμός λοιπόν ε, αφορά αυτού του είδους το σχεδιασμό. Το πρόβλημα για μας και έχω υποβάλει τροπολογίες 79, 81, 62 ε, σε συνεργασία και με τον συνάδελφο Χέιτεγκέντς και άλλους είναι το θέμα το οποίο ανέφερε ο κύριος Λάικφιντ προηγουμένως, δηλαδή το ύψος είναι πάρα πολύ, δεν είναι καθόλου πρακτικό να αλλάξει το ύψος. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε τη δουλειά που έχουμε ξεκινήσει. Υπάρχουν κάποιες ομάδες πίεσης και στο Ηνωμένο Βασίλειο και αλλού που είτε δεν μπορούν να διαβάσουν τις τροπολογίες είτε δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Σε μια τροπολογία εμείς λέμε ότι μπορούμε να δούμε ε, το ενδεχόμενο ε, μακρύτερων οχημάτων, αλλά εμείς δεν μπορούμε να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να, να, τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουν τα μακρύτερα ο, ο, οχήματα. και ανάλογα με τις ε, χώρες, ε, στη Σκανδιναβία ας πούμε, ξέρουμε ότι μπορούν ε, να βάλουν στους δρόμους τους πιο μακριά οχήματα. Τώρα, Ε, στην, ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, δεν είναι εύκολο να δεχτούμε για τους δικούς μας δρόμους αυτά τα μακριά, τα πολύ μακριά οχήματα, αλλά δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε να κινηθούν σε άλλους δρόμους. Το θέμα της οδικής ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό φυσικά και επίσης το θέμα της υποχρεωτικής αποδοχής οχημάτων που έχουν πάνω μηχανήματα που είναι αποδεκτά σε άλλες χώρες μέλη θα πρέπει να δούμε. Όσον αφορά ε, τις ε, κυρώσεις ε, και την τα μέτρα επιβολής του, του νόμου. Νομίζω ότι τα όσα αναφέρονται εδώ είναι ιδιαίτερα υποχρεωτικά και πολύ αναλυτικά. Νομίζω πάντως ότι μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο τελικό συμπέρασμα. Ε, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε κάποια υβριδικά ας πούμε, φορτηγά τα οποία είναι καλοσχεδιασμένα και τα οποία μπορούν να λύσουν ενδεχομένως το πρόβλημα του βάρους που μας απασχολεί. Νομίζω ότι θα πρέπει απλώς να σέβεται η μία χώρα την άλλη, να σεβαστούμε το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξουν και διμερείς συζητήσεις, αλλά χωρίς να προσπαθούμε να επιβάλλουμε κάτι στις ε, χώρες μέλη, να βρούμε ε, λύσεις ε, και, όσο, και, οι μεταφορείς να έχουν κάπως να διευκολυνθεί η ζωή τους έτσι ώστε να ε, μεταφέρονται με ικανοποιητικό τρόπο τα αγαθά τα οποία χρειαζόμαστε όλοι. Ο κύριος Ερτούκ, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστώ τον συγκητή για τη δουλειά του. Είναι δύσκολο βεβαίως να τοποθετηθεί καθνή ε, στο θέμα αυτό και να παραμένει μόνο στα αντικειμενικά στοιχεία, γιατί πάντα υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες και πάθη που αναδύονται. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, αγαπητοί φίλοι, για το πώς μπορεί κανείς να κάνει πολιτική για το συμφέρον των λόμπι. Και εδώ το βλέπω και το αιτιολογώ με τον τρόπο με τον οποίο έρχεται αυτή η πρόταση για τα liners, με μία μόνο επαγγελματική τάξη που μπορεί να κερδίσει από αυτήν την υπόθεση που είναι οι, ε, οι μεταφορτωτές των ε, εμπορευμάτων. Ούτε ο μεταφορέας, ούτε ο τελικός αποδέκτης, ούτε κανείς άλλος επωφελείται. Μόνο ο μεταφορτωτής μπορεί να μειώσει το κόστος του και έτσι να αυξήσει το κέρδος του από αυτό το μέτρο. Και γι' αυτό επιμένω ότι πρόκειται για ένα εσφαλμένο τρόπο να μιλήσουμε για διασυνοριακές μεταφορές. Διότι, για να μιλάμε καθαρά και να λέμε τα σίκα σίκα και το και τη σκάφη-σκάφη. Εδώ έχουμε να κάνουμε μια χαρακτηριστική περίπτωση σαλαμοποίηση τη νομοθεσία και το έχουμε γνωρίσει αυτό ήδη στη Γερμανία. Πολύ καλά μάλιστα το ξέρουμε. Και μάλιστα θα φτάσω να σα πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα έπρεπε πια να αντιδράσει και να προσπαθήσει αυτές τις ε, προσπάθειες που έχουν γίνει σε επιμέρους κράτη όπως η Γερμανία να τις αποτρέψει και να τις ανατρέψει γιατί έχουν οδηγήσει και σε καταστρατηγήσεις ε, της νομοθεσίας από τα εθνικά κράτη και συγκεκριμένα τη Γερμανία. Ε, έτσι λοιπόν ούτε γεωγραφικό περιορισμό έχει ούτε χρονικό περιορισμό έχει η Σαγάγη. Λέει ότι κάνει επιτόπου δοκιμές αλλά τελικά το μόνο που κάνει ότι νομιμοποιεί από την πίσω πόρτα αυτά τα Giga Liner, γιατί τίποτα άλλο δεν κάνει με αυτές τις υποτιθέμενες επιτόπου δοκιμές που θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξει πολύ πιο αυστηρά. Ένα παράδειγμα λοιπόν χαρακτηριστικό, όπως έλεγα, του τρόπου με τον οποίο τα λόμπι ε, εξασφαλίζουν ή τουλάχιστον βοηθάνε την ικανοποίηση των σφαιρώνων τους. Η κυρία Λίχτενμπέργκερ είπε πολλά, πολύ καθαρά. Μιλάμε για οι co και όλες αυτές τις θετικές πτυχές. Αλλά κανείς δεν μιλάει καθαρά για το γεγονός ότι αυτή η εξέλιξη και κάθε φορά αν χρειαστεί θα το επαναλαμβάνω, γιατί το πιστεύω και γιατί υπάρχουν και σοβαρές μελέτες πάνω σε αυτό, ότι η εισαγωγη του τέτοιου γίγα λάινερ θα έχει σαν αποτέλεσμα μεσοπρόθεσμα να έχουμε ακόμα λιγότερες ε, μεταφορές στους σιδηροδρόμους και ακόμη περισσότερες μεταφορές φορτίων στους δρόμους με αποτέλεσμα όπως είπε και η κυρία Λίκτινμπεργκερ, που το εξήγησε πάρα πολύ καλά ότι βεβαίω με τα αποτελέσματα αυτά που εξήγησε η κυρία και βεβαίω θέλουν τα λόμπι αυτό το μέτρο για το μέλλον γιατί τα συμφέρει. Το κόστος όμως θα πρέπει να το υποστεί η κοινωνία κάθε φορά, πράγμα το οποίο δεν δέχομαι. Δεν είναι λογικό περιβαλλοντικά. Και επεξήγηστε μου παρακαλώ Ποιο θα είναι εκείνο ο οποίο θα επιβαρυνθεί με το επιπλέον κόστο, όταν όλος, όταν ο κάθε μεταφορτωτή βγει από την αγορά και αρχίσει να λέει «Α, θέλω και εγώ αυτή τη δυνατότητα, θέλω και για μένα αυτή τη δυνατότητα» και έτσι θα έχουμε εν τέλει την ε, μεταφορά όλων των φορτίων ή των περισσότερων φορτίων από τους δρόμους μας και όχι από τους δρόμου. Απορρίπτω λοιπόν την πρόταση αυτή κατηγορηματικά. Ας κάνουν τα κράτη-μέλη ό,τι θέλουν, αλλά πάντως ακόμη και αυτές οι ε, δοκιμές επιτόπου όπως λέγονται πρέπει να ελεγχθούν και να περιοριστούν. Mr. Κύριε Higgins, ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Τώρα εδώ μιλούμε ουσιαστικά για το λόμπι των, ε, του κόμματος των Πρασίνων που θέλει να κάνει αυτή την ε, αντίθεση μεταξύ σιδηροδρόμου και οδικών μεταφορών. Ξέρουμε ότι, είμαστε, ότι είναι υπέρ των σιδηροδρόμων, αλλά δεν είναι και ρεαλιστές και βλέπουμε ότι υποβάλλουν τις ε, πλέον ε, γελίες ε, προτάσεις. Δεν ζουν στο δικό μας κόσμο λοιπόν, ζουν σε κάποιον άλλον κόσμο και έτσι ελπίζω να καταλήξουμε τουλάχιστον σε λογικούς συμβιβασμούς και συμβαστικές τροπολογίες. κύριος Πέτρης Σοβάνα που είπε εκ μέρους τον Σιωδών είπε ότι εδώ ουσιαστικά μιλάμε για μια φάρσα. Και το Βασίλειο και η Ιρλανδία είναι νησιωτικά έθνη και έχουμε επενδύσει τις υποδομές μας, ε, λαμβάνοντας αυτό υπόψη. Γιατί όμως η Επιτροπή Μεταφορών να έρθει τώρα τελευταία στιγμή και να μας πει να πει στα νησιωτικά ε, κράτη ότι δεν μπορούν να μεταφέρουν ε, ε, σε προϊόντα γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν σύνορα. Αυτό έρχεται απολύτω αντίθεση με τις τέσσερις ελευθερίες της Δηλαδή, με τα εμπορεύματα, τα πρόσωπα, τα κεφάλαια και τις υπηρεσίε και είμαι πεπισμένος ότι δεν συμμορφούνται ε, με τις συνθήκες. Το να περιορίζουμε δηλαδή το ε, εμπόριο μόνο βάσει των συνόρων που ανήκουν σε μια εποχή που έχει παρέλθει. Τώρα, για αυτά τα πολύ μεγάλα φορτηγά, αν δείτε στη Σουηδία, στη Φιλανδία και στις χώρες της Βαλτικής, τα χρειάζονται αυτά τα φορτηγά για, τη μεταφορά των προϊόντων τους. Δεν πρέπει να μπούμε σε μια τέτοια συζήτηση ε, όπου κάνουμε τη διάκριση ε, μεταξύ σιδηροδρόμου και οδικών μεταφορών. Λες και οδικές μεταφορές είναι κάτι που πρέπει να φοβόμαστε. Πρέπει να συνεπάρχουν αυτά τα δύο για το εμπόριο. Έχουμε κάνει πολλοί άριθμες ε, συζητήσεις με τον κύριο Σαβάραμα και άλλους βουλευτές και θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Φώστερ για τη στήριξή της. Ε, επί διαφόρων τροπολογιών. Γιατί τελικά εδώ μιλούμε για την αρχή της επικουρικότητας που είναι εξαιρετικά σημαντική σε ένα τέτοιο ζήτημα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ο κύριος Χίγγινς ε, υπενθύμησε τη συζήτηση που κάναμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τους ε, ταχογράφους και ε, τους αισθητήρε βάρους. Έχουμε παρατηρήσει ότι η λύση στην οποία καταλήξαμε δεν ήταν αρκετά όρημη και δεν είχαμε τη δυνατότητα να ε, βελτιώσουμε αυτό το στοιχείο στον κανονισμό για τους ψηφιακούς ταχογράφους. Όμως, σε ό,τι αφορά την πρόταση της Επιτροπής, ε, θεωρούμε ότι καλύτερο είναι να γίνει αυτό εδώ, σε αυτόν τον κανονισμό, για ε, το βάρος και το μέγεθος. Γι' αυτό και είχαμε κάποιες τροπολογίες, μέσω των οποίων επανεισήγαμε την χρήση των ευφυών ταχογράφων για τη μέτρηση της μάζας, και για την επαλήθευση του βάρους του φορτηγού. Νομίζω ότι πρόκειται για μια εφικτή πρόταση από τεχνική σκοπιά, παρότι η λύση δεν είναι αρκετά όρημη ακόμα. Όμως, ε, σε τεχνικό επίπεδο είναι εφικτό. Μια αυτόματη καταγραφή της ε, μάζας θα μας ε, επέτρεπε αυξημένα επίπεδα ασφάλεια στον δρόμο. Γι' αυτό και θα ήθελα να σα καλέσω να στηρίξετε αυτή την τροπολογία, γιατί ε, συνηγορεί προ αύξηση τη ασφάλεια. Ο κ. Καταρχά, όταν κάνει προτάσει νομοθετικέ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υποχρεωμένη να υποβάλει και τη σχετική ε, ε, ε, εκτίμηση επιπτώσεων, πράγμα το οποίο δεν έχει συμβεί εδώ πέρα, άρα βρίσκεται σε παραβίαση συνθήκης, έχουν περάσει ένα, δύο, τρία χρόνια και δεν υπάρχει καμιά έρευνα και πρέπει αυτό να αποτελέσει προϋπόθεση πριν να εισεχθεί οποιοδήποτε άλλο, οποιοδήποτε άλλο νομοθέτημα. Υπάρχει που μας λένε ότι το 35% των ε, μεταφορών έχουν, φορτίων έχουν περάσει των επιμέρους μεταφορών φορτίων έχουν περάσει από το σιδηρόδρομο στις οδούς και, θα, και συμβαίνει και το ίδιο και με τις συνδυασμένες μεταφορές προς το 50%. Ε, θα είναι ακόμα πιο έντονο αυτό το φαινόμενο ε, και ουσιαστικά έχουμε με αυτόν τον τρόπο ε, παραβεί τους όρους της Λευκής Βίβλου. Δεν εφαρμόζονται λοιπόν οι στόχοι της που έχουμε ορίσει με την Λευκή Βίβλο και υπεύθυνοι γι' αυτό δεν είναι η πράσινοι όπως λέτε, αλλά εσείς οι οποίοι προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε μόνο τα λόμπι. Ο ανταγωνισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται, υπήρξε μια παρέκκληση για τη Σουηδία και τη Φιλανδία που είχαν ήδη τα πολύ βαρέα οχήματα, τα πολύ μακρά οχήματα και το ανεχόμαστε γιατί εδώ και καιρό χρησιμοποιούν αυτά τα οχήματα, όλα τα άλλα απαγορεύονται. Όμως πριν από τέσσερα χρόνια ο επίτροπο Κάλλα υιοθέτησε, ε, με, σε μια δική μου ερώτηση, κατηγορηματικά την διαθέση και δύο χρόνια μετά λέει α, όχι δεν ισχύει αυτό. Λοιπόν δεν γίνεται, δεν επιτρέπεται και επίση υπάρχουν πολλέ εκδηλώσει από την Daimler την εταιρεία που, κατασκευάζει αυτά τα μεγάλα φορτηγά και που είναι κατηγορηματικά κατά της χρήσης του γιατί λέει ότι θα υπάρχουν πολύ σοβαρές συνέπειες. Δεν του συμφέρει δηλαδή ένα ή δύο φορτηγά να αξιοποιηθούν. Αυτοί και και οι ίδιοι δηλαδή θεωρούν ότι δεν είναι συμφέρουσα η χρήση των μεγάλων αυτών φορτηγών για τις μεταφορές ε, γιατί ε, πάνε μένα, αλλά πρέπει μετά να βρουν φορτίο για να γυρίσουν και δεν είναι συμφέρον να ταξιδεύουν πίσω άδεια. Το ίδιο βλέπουμε στο Λίμπεκ μια ε, γέφυρα πρέπει να κλείσει γιατί δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί από απλά ε, οχήματα έχει πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή δεν υπάρχουν εν γέννη υποδομές, γιατί το βλέπουμε παντού αυτό και κάποιοι που θέλουν να οξύνουν αυτό το φαινόμενο, ε, αυτά τα monster trucks, τι να σας πω, βάλτε τα πάνω σε όλους τους δρόμους της Ευρώπης να καταστραφεί κάθε γέφυρα που μας έχει μείνει. Για δε τα ουσίδηροδρόμους, 30 δισεκατομμύρια μόνο για την εξυγίανση των γεφυρών και δεν μιλάω για το οδικό δίκτυο, ε, θα χρειαστεί για να προχωρήσει αυτό. Για τρία χρόνια τα λόμπι των φορτηγών στη Γερμανία τάσσονταν κατά των ε, τεράστιων αυτών φορτηγών. Τον ένα λόγο, μάλιστα τον παρουσίασε στην ε, Ομοσπονδιακή Βουλή ο Επίτροπος Κάλλας, διότι είναι πάρα πολλές θέσεις εργασίας στα ε, μικρότερα φορτηγά. Ένας αυτά τα monster trucks, αντί για τρεις-πέντε οδηγούς θα χρειάζεται μόνο ένας. Άρα επιδεινώνονται τα προβλήματα και στην απασχόληση. Πολύ σημαντικό αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να κατευθυνθούμε προς άλλες λύσεις. Ε, και πιο οικολογικές και πιο οικονομικές, ε, πράγμα το οποίο δεν ισχύει με τα γίγα, δεν ισχύει με τα γίγα τραξ. Σε μία κρόση πρόσφατα στη Βορειοερνωνία Βεσφαλία, στο τοπικό κοινό βούλιο, άκουσα ότι άπαξ και επιτραπεί η κυκλοφορία αυτών των μεγάλων φορτηγών σε ένα σημείο, τότε αμέσως θα προχωρήσει η πίεση και μάλιστα από το, τον άστο 60 τόνων θα πάει στα 80 και μετά όλο και παραπάνω. Αυτή είναι η τακτική που ακολουθείτε. Μπορεί να γνωρίζετε οι Ολλανδοί και οι Βέλγοι ότι ε, μια μέθοδος ε, σταδιακής πίεσης μπορεί να φέρνει αποτελέσματα, αλλά σας διαβεβαιώ ότι η Βόρεια Αρνανία Βεσταλία θα αρνηθεί μέχρι τελευταία. γιατί εσάς μόνο η, η γραμμή Rotterdam Anversas δεν μπορεί να σας είναι χρήσιμη αν δεν μπορείτε να περάσετε μέσα από τη Γερμανία. Εξού και δεν συζητάτε άλλα ζητήματα. Οι υποδομές λοιπόν θα χρειαστεί να επεκταθούν, θα χρειαστεί να υποστηριχθούν, πράγμα το οποίο σημαίνει και ιδιωτικοποίηση και λύσεις που θα αποβούν χρήσιμες μόνο για ορισμένε επιχειρήσεις και μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον. Και γι' αυτό το ζητάτε εσείς, ε, ε, γι' αυτό εμείς είμαστε κατά των ε, μεγάλων αυτών φορτηγών και δεν είμαστε κατά των πάντων όπως λέτε γιατί υπάρχουν πολλά άλλα θέματα στα οποία υποστήριξαμε τις εξελίξεις. Εμείς είμαστε πάντα υπέρ, τώρα ανανεώσιμος, ναι με συγχωρείτε Πρόεδρε που ήμουν μακριά από το μικρόφωνο, ε, ήμασταν πάντα υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και γι' αυτό θέλω να δω πρώτον μια ε, μελέτη επιπτώσεων πριν από την νομοθεσία. Και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστώ. Να θυμίσω απλώς στου συναδέλφου ότι εγώ δίνω το λόγο, η Προεδρία δίνει το λόγο. Δύο λόγια να πω κι εγώ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά το ζήτημα Ηνωμένου Βασιλείου Ιρλανδίας, το γεγονός ότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία χρόνια παρα, ε, δρούν παρανόμως, ε, δεν σημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Επίσης, το ζήτημα της ασφάλειας είναι πολύ σημαντικό. Εάν χάσουμε αυτό το θέμα της ασφάλειας, τότε θα μπούμε σε μια τελείωτη σειρά οικονομικών εμπορικών ε, ε, συζητήσεων. Γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ με τα πιο μακριά οχήματα φορτηγά. Μπορεί κανείς βέβαια να έχει μακρύτερα ε, φορτηγά που ζυγίζουν το ίδιο με τα υπάρχοντα ή ε, που ζυγίζουν και πιο λίγο. Το θέμα είναι το βάρος βέβαια, να είμαστε ε, ειλικρινείς και να μιλήσουμε ξεκάθαρα, να πούμε ότι μιλάμε για βαρύτερα οχήματα. Όταν αναφερόμαστε σε οικονομικά πλεονεκτήματα. Βεβαίως, καταλαβαίνω ποια είναι τα πλεονεκτήματα. Γι' αυτό είναι πολλοί αυτοί που ε, ταράζονται και το θέλουν αυτό. Το θέμα είναι ε, ποιος είναι αυτός που θα πληρώσει τελικά αυτή τη διευκόλυνση, ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό, ο φορολογούμενος. Δηλαδή πάλι οι ίδιοι θα πληρώσουν την υποδομή αυτή. Πριν από χρόνια όταν ήρθα στο κοινοβούλιο ε, είχε ξεκινήσει μια συζήτηση για τις μεταφορές και πάλι συζητούσαμε με, τα ίδια, με τους ίδιους όρους. Τι να σας πω τώρα, και όλη αυτή η συζήτηση ε, με και όλο αυτό το, ε, ζήτημα με τους ε, φορτηγατζίδες οι οποίοι πάνε και πέφτουν πάνω στις γέφυρες του σιδηροδρόμου έχουν κάτι. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο μακρύ, πόσο φαρδί, πόσο βαρύ είναι, αλλά είναι πρόβλημα όλα αυτά τα φορτηγά τα οποία χώνουν τη μύτη τους στη δουλειά των σιδηροδρόμων και προκαλούν πολύ μεγάλα προβλήματα. Κύριε Ισηγητά, κύριε Λάιτφρεντ, πολύ με απογοητεύσατε με την έκθεσή σας, γιατί νομίζω ότι είσαστε πολύ μετριοπαθείς. Κυρίως όσον αφορά αυτό που ανέφερα μόλις. Αλλά σε ένα πνεύμα συνένεσης ε, είπα να συμφωνήσω με την ε, άποψη του κυρίου Φράιντ. Ε, εγώ σαν, σαν όχι σαν πρόεδρος αλλά αντιτίθεμαι στα πιο φαρδιά οχήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακούσαμε 16-17 παρεμβάσεις σήμερα. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι κατά την άποψή μου στηρίζουν την αναθεώρηση κυρίως, κυρίως όταν ε, μιλάμε για, πρασιν, για πιο οικολογικά ας πούμε και πιο ε, καθαρά ε, φορτηγά. Είναι 300 και, πάνω από 350 οι τροπολογίες, όσες και οι μέρες του χρόνου. Για να δούμε πώς μπορούμε να τα βολέψουμε τα πράγματα. Να πω δύο λόγια πρώτα απ' όλα σχετικά με τις τροπολογίες αυτές. Μερικές ε, βελτιώνουν ε, την πρότασή μας ας πούμε ε, όσον αφορά την, το επιπλέον βάρος για εναλλακτικά συστήματα προώθησης. Αυτό τα καλαδεχόμαστε αλλά μας εκπλήσουν τροπολογίες οι οποίες ε, θέλουν να διαγράψουν την πρόταση. Εδώ έχουμε μια πρόταση η οποία σύμφωνα και με την ε, αξιολόγηση αντικτύπου που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του προηγούμενου χρόνου ε, μπορεί να μειώσουν τις εκπομπές των των φορτηγών κατά 10% χωρίς να αλλάξει καθόλου η φορτωτική τους ικανότητα. Επίσης βελτιώνουν την ασφάλεια ε, και αυτό είναι καλό για όλη την κοινωνία γιατί βελτιώνει την ε, ορατότητα του οδηγού. Η Κομισιόν βεβαίως δεν μπορεί να δεχτεί και τροπολογίες οι οποίες αμφισβητούν ε, τον στόχο της οδηγία ή ας πούμε αυτή που αναφέρεται σε μείωση του, όγκους, του, του μήκους των ρημουλκωμένων. και ξέρουμε ότι το, το μήκος το οποίο μπορούμε να δεχτούμε είναι ε, το πολύ, ε, αντί του 50 που έχουμε προτείνει, 200 σαντιμέτρα. Επίσης, ε, οι προθεσμίες, ορισμένες τροπολογίες ζητούν επιπλέον καθυστέρηση αλλά ε, κοιτάξτε, αυτό το θεωρώ λυπηρό. Ε, η Ευρωπαϊκή Αυτοκινητοβιομηχανία, ίσω όχι στο σύνολό τη, αλλά πάντω έχει κάνει μεγάλε ε, επενδύσει. Και τώρα του λέμε περιμένετε, δεν πειράζει που κάνετε την επένδυση, περιμένετε και θα δούμε. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τέτοιε τροπολογίε. Η πρόταση αυτή αφορά οχήματα τα οποία θα είναι πιο καθαρά, πιο φιλικά προς το περιβάλλον, πιο αποτελεσματικά, πιο ελαφριά. Και στην ουσία ε, δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί ότι ε, μιλάμε για πιο βαριά οχήματα και για πιο μακριά οχήματα. Αντιθέτως ε, μιλάμε για μικρότερες εκπομπές, για λιγότερους ρήπους, για καθαρότερα φορτηγά. Κοιτάξτε λίγο, σας το ξαναλέω, την μελέτη αντικτύπου την οποία έχει δημοσιοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τίποτα δεν υπάρχει στην ε, ε, οδηγία ε, που να απαγορεύει την διακίνηση αυτών των, ανθρω... αυτών των τροποποιημένων φορτηγών μεταξύ δύο χωρών που επιτρέπουν την κυκλοφορία τους. Και νομίζω ότι κατά αυτήν την έννοια γνωμοδότησε και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι είναι λίγο συγκινησιακή αυτή η συζήτηση που γίνεται εδώ. Πριν από χρόνια όταν ξεκίνησε η συζήτηση αυτή ε, νομίζω ότι πάλι είχαμε την ίδια ε, έτσι, συγκινησιακή αντιμετώπιση η οποία μας έβγαζε λίγο από τον στόχο της ε, συζήτησης. Επομένως, καμία χώρα μέλος δεν μπορεί να υποχρεωθεί να δεχτεί πιο μακριά οχήματα, αυτό είναι σαφές. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια των μακριτέρων οχημάτων. Οι ίδιοι εμπλεκόμενοι αναφέρονται ε, σε υψηλό κόστος προσαρμογής των υποδομών. Αυτό θα πρέπει να το δούμε προσεκτικά. Όσον αφορά την ασφάλεια, αυτά που ξέρουμε από πραγματικά ε, ε, πειράματα που έγιναν σε χώρες μέλη είναι ότι η χρήση μακριτέρων οχημάτων δεν έχουν περισσότερα ατυχήματα από τα στάνταρτ. Ίσως γιατί οι οδηγοί είναι καλύτερα εκπαιδευμένοι, ίσως γιατί κάνουν συγκεκριμένες διαδρομές, δεν το γνωρίζουμε. Ε, θα πρέπει κανείς ε, να διαβάσει ε, τις, τα αποτελέσματα των δοκιμών στη Δανία και στην Ολλανδία. Απ' την άλλη πρέπει να δούμε ποια είναι η περιοχή, ποια είναι η κατάσταση στις αστικές περιοχές. Στην Γαλλία υπάρχουν ήδη λεωφορεία 24 μέτρων μήκους ε, και δεν γίνεται λόγος γι' αυτό για, για αυτά τα λεωφορεία και μιλάμε διαρκώς για αυτά τα μακρύτερα φορτηγά τα οποία θα κυκλοφορούν ενδεχομένως σε αστικές περιοχές. Επίσης, από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιες ιδέες σχετικά με τους ε, διαδρόμους. Ε, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να το δούμε η προσέγγιση για αυτού του είδους ε, τα ε, φορτηγά μπορούν να διατηρήσουν τα δικαιώματα των κρατών και να ε, προωθήσουν τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Και βεβαίως μιλάμε για οχήματα τα οποία θα κυκλοφορούν μόνο με καλά, κατάλληλα εκπαιδευμένους οδηγούς και που θα κυκλοφορούν μονάχα σε αυτοκινητοδρόμους που έχουν προβλεφθεί για τούτου είδους ε, τα οχήματα. Πάντως ε, πρέπει να πω και να αναγνωρίσω ότι ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε πιο αποτελεσματικά, ενεργειακά, ε, καθαρά και ασφαλή οχήματα και νομίζω μέσω της οδηγίας αυτής συνδυάζονται όλοι αυτοί οι στόχοι. Ξέρω ότι οι φίλοι μου από αυτή την πλευρά του Κοινοβουλίου δεν συμφωνούν, αλλά παρόλα αυτά ε, πρέπει να τους πείσω και πρέπει να τους το ξαναπώ ότι εδώ μιλάμε για πιο καθαρά, πιο πράσινα οχήματα, τα οποία και πιο ασφαλή μπορεί να είναι και πιο αποτελεσματικά. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα μόνο να πω ότι ε, ο εκπρόσωπος, ο συνάδελφος από το ECR... Ε, χαιρέτησε και χειροκρότησε τον συνάδελφο από την Κομισιόν. Ελπίζω να το κάνει το ίδιο και για άλλα ζητήματα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο για τον κύριο Μπένιον. Νομίζω ήθελα να διευκρινίσουμε αν η Επιτροπή θα θέσει όρια στα ε, flaps ε, και στα caps. Είναι μια νέα προσέγγιση, δηλαδή που δεν πρέπει να ορίζουμε πώς, τι μορφή θα πρέπει να έχει ε, το φορτηγό, αλλά να προσδιορίσουμε τι πρέπει να κάνει αυτό το, το φορτηγό. Για τις μέγιστες διαστάσεις θέλουμε να έχουμε ε, βασικά κριτήρια αποδοτικότητας, ε, το οποίο έχει μεγαλύτερη ευελιξία για το μέλλον, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν η τεχνολογία, πώς θα εξελιχθεί η τεχνολογία. Γι' αυτό δεν έχουμε εξειδικευμένε προδιαγραφέ και γι' αυτό μιλήσαμε για τα flaps. Γιατί έλεγχη κάθε 2.000 χιλιόμετρα. Βρήκαμε ότι το υπερβολικό βάρο ε, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ε, στο δικό δίκτυο και δεν λειτουργούν οι έλεγχοι. Είναι πρόβλημα για τι υποδομέ και για την οδική ασφάλεια και θέλουμε να βοηθήσουμε τα κρατημέλη να προστατεύσουν ε, το δικό τους δίκτυο, να αυξήσουν την ασφάλεια στο δρόμο. Γι' αυτό και έχουμε θέσει τα 2.000 χιλιόμετρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε τα φορτηγά. Αντιθέτως, θέλουμε να έχουμε τεχνικές λύσεις που έτσι θα έχουμε ε, την τζίγηση εν κινήσει. Με αισθητήρε ε, ε, βάρους μπορούμε να εντοπίσουμε και να ζυγίσουμε το φορτηγό χωρίς να το σταματήσουμε και αν εντοπιστεί πρόβλημα τότε το σταματάμε. Αυτά ήθελα να πω. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Mr. Κύριος Λάιτφριντ. Αξιότιμα μέλη, αρκετά, αρκετές κατηγορίες ακούσαμε δεξιά και αριστερά. Παρακαλώ μην κατηγορείτε έτσι ελεύθερα. Κύριος Λάιτφριντ. Ναι, κατανοώ ο πρόεδρο ότι θέλετε να περισπιστείτε τον εαυτό σας, αλλά το να φωνάζει ο ένας στον άλλον κατηγορίες, να λέγεται τη έρθουσα, δεν ε, ωφελεί. Κυρία Λίχτεμπεργκερ, δεν επικρίνω τον έναν αντί για τον άλλον. Ακούσατε τη δική μου προσωπική άποψη. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Λάιτφιντ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τρίτη και καλύτερη παρέμβαση. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μάισνερ γιατί κατάφερα να, και σημείωσε και η ίδια ότι κατάφερα να μείνω πάρα πολύ ήρεμος και ψύχρεμος. Πραγματικά προσπάθησα να το κάνω. Και νόμιζα ότι όλοι αυτό πρέπει να κάνουμε, ειδικά ω εισηγητές, αν θέλουμε να έχουμε και αποτελέσματα. Αλλά έχασα κάπως την ψυχραιμία μου, ιδίως ακούγοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν η ΠΕΤΡΟΠΗ θέλει να μας ε, κάνει διδάγματα για τη ζωή, ας ρωτήσει τους Ευρωπαίους πολίτες ποια είναι η δική τους γνώμη για την πραγματική ζωή εκεί έξω. Και ας μην ε, προσποιούμεθα ο ένας μπροστά στον άλλον. Υπάρχουν ε, μερικά σημεία που θα πρέπει να θίξω. Εάν θέλει ο κύριος Κάλλας να υπάρξει νόμος που αφορά τις χαμηλότερε εκπομπές και μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος, μεγαλύτερη ασφάλεια στο, στο οδικό δίκτυο, θα πρέπει να κάνει νομοθεσία ακριβώς για αυτό το σκοπό και όχι να ψάχνει να το βρει όλο αυτό αλλού και μετά να διαρωτάτε γιατί συζητούμε κάτι άλλο και να μην ακολουθεί μόνο τα λόμπι. Και άλλοι το είπαν αυτό, ότι είναι υπερβολικό κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επιστρέφω και πάλι στον ψύχρωμο εαυτό μου. Και τώρα θα ήθελα να αναφέρω ε, σημεία που έθιξαν συνάδελφοι. Ο κύριος Μαντάλεν είπε κάτι το οποίο με εξέπληξε ιδιαίτερος. Είπε ότι αυτά τα mega ή τα eco φαντάζομαι ότι μπορεί να μην είναι καλά. Αλλά δεν υπάρχουν τροπολογίες που να αντιστοιχούν σε αυτή την παρατήρηση. Γιατί κυρία Λίχτεμπεργκερ και την ηλεκτρονική όθηση δεν είναι ότι αυτά τα φορτηγά αντλούν ηλεκτρική ενέργεια από εξωτερικές πηγές. Την παράγουν εν κινήσει. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Όμως ε, θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό και για τα συνδροδρομικά δίκτυα όταν ε, μιλάμε για περιβαλλοντικά συστήματα. Έτσι έχουν τα πράγματα λοιπόν. Ουσιαστικά πρέπει να βρούμε μια λύση που θα είναι προς όφελος της Επιτροπής. Θα έχουμε νόμο που θα αφορά τις εκπομπές, ε, την ασφάλεια και την οικολογία. Οτιδήποτε άλλο έχει τύχη προετοιμασίας. Και αν θεωρεί η Επιτροπή ότι χρειάζεται αξιολόγηση δικτύπου... Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από πυρογνώμονε ε, να το παρουσιάσει, γιατί η Κομισιόν ήθελε εξολόγηση τύπου. Τέλο πάντων, οι απόψει μα διαφέρουν από αυτού. Και τέλος, να καλέσω τον ε, κύριο Higgins ε, να επανεξετάσει ένα θέμα που ανέφερε και ο Πρόεδρος. Δεν ήταν πρόταση της Κομισιόν που ήθελε να απαγορεύσει κάτι τέτοιο στη Βορειοελλανδία. Ούτε ο εισηγητής ήθελε κάτι τέτοιο. Τώρα κατά πόσο αυτή η πρακτική που ισχύει εδώ και χρόνια είναι παράνομη ε, και θέλω το θέσει αυτό κατά μέρος η Επιτροπή και να βρει μια λογική λύση για το μέλλον θα δούμε αν μπορεί να συνεχιστεί αυτό για χρόνια ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Φεβρουαρίου, ενδιαφέρουσα θα γίνει αυτή η ψηφοφορία σίγουρα και στην Ολομέλεια ε, προγραμματίζεται για τον Απρίλιο, αλλά δεν ξέρουμε ακόμα αν θα γίνει τότε, γιατί βεβαίως ε, όλοι θα θέλουν να ψηφιστούν οι εκθέσεις τους τον Απρίλιο. Λοιπόν, 11 Φεβρουαρίου η ψηφοφορία. Σας ευχαριστώ για την ε, πολύ αυτή ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να υπενθυμίσω στα μέλη ότι η επόμενη συνεδρία θα γίνει την 5η, συγγνώμη, 5η λοιπόν 30 Ιανουαρίου στις 9. Να ευχαριστήσω και τους διερμηνείς. Καλό απόγευμα σε όλους.